Uh, well, good morning, everybody. We just, um, I just heard the news that our rapporteur. Καλημέρα σας. Δυστυχώς ο εισηγητής μας ασθενεί σήμερα το πρωί. Ο κύριος Φάντ όμως θα το παρουσιάσει. Αντί του Παύλου Αρίας Ετσεβερία, θα να αρχίσω τη συζήτηση για τη σημερινή μας ε, ημερήσια διάταξη. Συγγνώμη, αργήσαμε λίγο. Ναι. Κάτι το οποίο βέβαια συμβαίνει συχνά αυτέ τι μέρες. Τέλος πάντων, ε, 10 θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Πολύ σημαντικές ψηφοφορίες. Παρ' όλα αυτά πιστεύω θα προλάβουμε να συζητήσουμε αυτή την έκθεση, την πολύ σημαντική, του κυρίου Αρίας μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατόπιν εκθέσεως στρατηγικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέκυψε από πολλές ε, συζητήσεις γύρω από την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως επίσης και τη δουλειά της δικής μας Επιτροπής στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, που ο κύριος Αρίας τη οποία ο κύριος Αρίας ηγείται μαζί με άλλους συναδέλφους. Αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μας στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα δούμε τι νομοθετική δράση θα αποφασιστεί στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία και θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Αρίας είναι ο εισηγητής μας. Η κυρία Σάλοβα είναι εδώ, σκιώδης εισηγήτρια. Ασχολείται και με την πρόταση e-call ε, και συμμετέχει και στην Επιτροπή με τα μεταφορών. Ε, Ρούιλε και Κρόιτσμαν είναι εδώ. Όχι, η κυρία Ρούιλε δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κρόιτσμαν είναι εδώ. Ο κύριος Πέρνερστινγκ είναι εδώ. Α, δεν είναι. Α, εσείς τον εκπροσωπείτε. Καλώς. Και είναι εδώ και εκπρόσωποι της Γενικής ε, Διεύθυνσης ε, Αγορών. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σφάμπεκ, μέρους του εισηγητή να μας πει την άποψή του για τις έξι τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι εμείς άρχισαν πολύ νωρίτερα από άλλες επιτροπές. Η ΕΚΟΝ καμία σχέση, ακόμα δεν έχει αρχίσει. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά ε, δεν πειράζει. Ε, καταφέραμε επιτέλους και για τις υπηρεσίες πληρωμών να βρούμε μια συμβαστική πρόταση προς τη σωστή κατεύθυνση για την ψηφοφορία. Και ένα τρίτο που έχω να πω, πραγματι ο συνάδελφος Παμπλο Άριας, που ε, έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ προσυρωμένα και με μεγάλη πειθαρχία σε αυτό το θέμα, δυστυχώς σήμερα χρειάζεται να νοσηλευτεί στη Μαδρίτη, είχε χειρουργηθεί στο γόνατο και βρέθηκε και άλλη υποκείμενη ε, βλάβη που δεν την είχαν ανακαλύψει και πρέπει να είναι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ας έρθουμε στις ε, λεπτομέρειες. Στα αγγλικά, κύριε Σουάμπ, για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητή ε, χαίρεται για τη συνεργασία που είχε με το σκιώδη εισηγητή και τη γενική συνένεση με την, στην οποία κατέληξαν ε, στις βασικούς τομείς του θέματος αυτού. Το είδαμε αυτό και στη Γενική Ανταλλαγή Απόψεων στις 25 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Αρίας είναι της απόψεως ότι περισσότερες τροπολογίες είναι πολύ θετικές και συμμετέχουν στη βελτίωση του, ε, ε του κειμένου, του, κύριο Κρόιτσμαν, την κυρία Ρούλερ, τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον, την κυρία Σαβίνη θα ήθελε να ευχαριστήσει μεταξύ άλλων. Ε, βλέπω ότι επιστρέφει ο κύριος Τριανταφυλλίδης και χαίρομαι γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ για το θέμα της ε, οδηγίας δικαιωμάτων καταναλωτών. Τι άλλο μου ζήτησε να κάνω ο Πρώτον, υπάρχουν πολλές τροπολογίες που εστιάζουν στις ε, συνθήκες εργασίας στην αγορά παράδοσης δεμάτων ε, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης και στη Γερμανία. Θέλει λοιπόν ο κύριος Αρίας να επιμείνουμε σε σωστές συνθήκες εργασίας βάσει της εθνικής νομοθεσίας με προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο αναφέρεται στις τροπολογίες. Πρέπει όμως να μην μας διαφεύγει ότι το θέμα του τρέχοντος ε, φακέλου είναι να ολοκληρώσει την αγορά παράδοσης δεμάτων και ο στόχος είναι μία ψηφιακή οικονομία, κάτι το οποίο έχουμε ψηφίσει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και πρέπει συνεπώς να επικεντρωθούμε ε, στην ε, ε, προσπάθεια να βελτιώσουμε την αγορά αυτή χωρίς όμως να μειώσουμε τις συνθήκες, την ποιότητα των συνθήκων εργασίας στον τομέα αυτών. Επίσης ο κύριος Αρίας παρατηρεί ότι σε κάποιους τόπους δεν συμφωνεί με την, ε, με την ε, προσθήκη ενός υπότιτλου στο 18. Πιστεύει, να, πιστεύει ότι είναι καλύτερα να διατηρηθεί ε, ο τίτλος ως έχει. Συμφωνεί όμως με τις 19, 20 και 21 για τα αξιόπιστα, για τους αξιόπιστους ιστοτόπους. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες όσον αφορά τη δημιουργία ενός σήματος εμπιστοσύνης για το ηλεκτρονικό εμπόριο και αυτό είναι κάτι για το οποίο ο Παύλο Αρίας ε, στη προσπάθεια του, από τότε που ξεκίνησε την προσπάθεια ε, εξέτασης αυτού του θέματος, ε, πάντοτε συμφωνούσε και ελπίζει ότι η τροπολογία 16 που είναι μια συνένεση μεταξύ όλων των ε, τροπολογιών διαφόρων πολιτικών ομάδων ε, ε, μπορεί να διατηρηθεί. Συμφωνεί με τις τροπολογίες του κυρίου Κορέα Ντεκάμπος για τα διάφορα θέματα που αφορούν αυτές, όπως επίσης και των κύριων Μπίλαν και Κρόιτσμαν. Και η δική μου ακόμα τροπολογία 54 τον βρίσκει σύμφωνο, με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Ο κύριος Αρίας λοιπόν με πολύ χαρά θα συνεργαστεί περαιτέρω με, την, ε, με τους συναδέλφους ε, για τη συνέχιση του, ε, του θέματος αυτού και λυπάται πολύ που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ανάρρωση ευχόμαστε στον κύριο Παύλο Αρίας. Ξέρω ότι έχει πολύ καιρό πρόβλημα, μήνες τώρα με το γονατό του. Ελπίζω να περάσει τώρα με την εγχείρηση. Κυρία Σενέλοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρόκειται για μια γνωμοδότηση ε, στην ε, Επιτροπή Μεταφορών ε, και πρέπει να πάω και εκεί. Εν πάση θέλω να σα πω ότι έχουμε ξανακάνει ανταλλαγή απόψεων και ο εισηγητή, ο κύριο Άρια, κατά την άποψή μα, ακολουθεί καλή ε, οδό και στι τροπολογίε μα προσπαθήσαμε Ε, να ε, επικεντρωθούμε σε κάποια θέματα που χρειάζονται μεγαλύτερη εστίαση. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ συντομία σε μερικές από τις τροπολογίες. Η πρώτη θεματική ενότητα έχει να κάνει με την αγορά στην Ευρώπη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παράδοση είναι ευκαιρία και για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών ή των παροχωμένων υπηρεσιών και θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, τονωθεί η εμπιστοσύνη. Πρέπει να υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία για να ε, οριστούν ελάχιστες προδιαγραφές και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος θα δίνει την πιστοποίηση και την έγκριση. Θα είναι μια κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία ή ένα χώρα μέλος. Επίσης, ε, και πάντα προς το συμφέρον των καταναλωτών, οι πληροφορίες που θα δίνονται ε, θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και θα πρέπει να αφορούν ε, και την παρακολούθηση ε, τη αποστολής, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, να μπορεί ο καταναλωτή ηλεκτρονικά να το παρακολουθεί. Ε, σήμερα αυτά γίνονται πάρα πολύ κωδικοποιημένα και είναι πολύ δύσκολο για τους ε, καταναλωτέ να παρακολουθούν την πορεία του δέματο. Επίσης, κάτι άλλο που υπόθηκε στην προηγούμενη συζήτηση, στις προηγούμενες συζητήσεις είναι η βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψης και η ε, κάλυψε και η ταχεία παράδοση σε απομακρυσμένες αραιοκατοικημένες περιοχές στην Ήπεθρο, σε πόλεις και χωριά. Ε, επίσης, οι διαδικτυακές πύλες ε, να μπορούν να είναι συγκρίσιμες γιατί όλο και περισσότεροι καταναλωτές ανατρέχουν σε αυτές τις ιστοσελίδες και συγκρίνουν τιμές, προθεσμίες, παράδοσης και άλλα τέτοια στοιχεία. Αλλά ε, αυτά όλα δεν είναι πάντα με την απαραίτητη διαφάνεια σχεδιασμένα στο διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, αξιοπιστία και ενημέρωση, αλλά κυρίως ανεξαρτησία προς όφελος πάντα των καταναλωτών. Και ε, ένα άλλο θέμα επίσης σημαντικό είναι κάτι που επίσης έχω ξαναπεί σε προηγούμενες συζητήσεις μας. Και αυτό είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ολοκληρωμένης αγοράς για την αποστολή ε, δεμάτων. Και εδώ ε, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι καλές συνθήκες εργασίας και χαίρομαι που το λαμβάνει αυτό ε, υπόψη του και μια σειρά συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες. Πολλές φορές βλέπουμε καταχρήσεις ή παραβιάσεις των θυστικών εργασίας. Οι εργαζόμενοι έχουν επισφαλή συμβόλαια, συμβάσεις ορισμένου χρόνου με κακές συνθήκες και κριτήρια που δεν πληρούνται πάντα και όλα αυτά δεν συνάδουν με αξιοπρεπείς μισθούς ούτε αξιοπρεπή εργασία και στη συνέχεια αυτό έχει και αρνητική επίπτωση ε, στο ίδιο το αντικείμενο, στην αποστολή και παράδοση. Μας ενδιαφέρει πολύ η κατάρτιση των εργαζομένων. για να υπάρχει ακριβώ μια ενιαία αγορά ολοκληρωμένη και συγκρίσιμη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά προς το παρόν. Χαίρομαι που θα το ξαναπούμε με τον εισηγητή, τον κύριο Άριας και ε, που βρήκαμε ένα καλό δρόμο να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προσωπικά έχω κάνει λίγες τροπολογίες γιατί ε, με ικανοποίησε πολύ το σχέδιο έκθεση του κύριου Άρια. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερη ενημέρωση για τις ε, παρεχόμενες υπηρεσίες στο μέλλον. Θα πρέπει να είναι πιο εύκολο στο διαδίκτυο κανείς να συγκρίνει τις διάφορες προσφορές. Εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν κοινού δείκτες ε, για να αξιολογούμε την ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης ε, προϊόντων. Ε, συνεργάζονται ε, οι αρμόδιοι με τις ενός καταναλωτών. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ε, μεταξύ των μεγάλων κολοσσών όπως είναι η Amazon και των μικρών εταιριών που στέλνουν δέματα ε, ως προς το κόστος ε, αποστολής και παράδοσης. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η συνένωση ας πούμε μικρών εμπόρων σε ενώσεις που θα παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες για να αυξηθεί το δυναμικό τους. Επίσης, ε, έχουμε και ορισμένες ε, υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού το ταχυδρομείο και κάποιες ε, εταιρείες ταχυμεταφορών και παράδοσης δεμάτων, courier δηλαδή. Αυτά όλα μπορούν να συνδυαστούν κάλλιστα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ε, τόλμησα να αναφερθώ σε δύο νομοθετήματα που θα βοηθήσουν και θα δώσουν φτερά στην ολοκλήρωση ε, μια ενιαία δήλωση ΦΠΑ και ε, ένα ε, εμπορικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προαιρετικό όμως. Υποστηρίζω την πρόταση ε, του εισηγητού να εκπονηθεί ένα ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μπορεί να έχει, μην έχει άμεση σχέση αυτό με την παράδοση δεμάτων, αλλά είναι σχετικό. Προσοχή όμως αυτό το εμπορικό σήμα να μην το υπερφορτώσουμε, γιατί θέλουν προφανώς πολλοί εμποροί να το χρησιμοποιούν. Ε, θα πρέπει ε, να εστιάσουμε στα κριτήρια που είναι σημαντικά για του καταναλωτέ, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η τήρησή τους θα πρέπει να απαντά σε κριτήρια εφορίας, ε, όχι όμως οικολογικά και τέτοιου τύπου, διότι δεν έχουν σχέση πάρα πολύ με το συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι πολύ ε, δύσκολος ο έλεγχος όταν είναι πολύ περίπλοκα τα κριτήρια. Ε, κανείς δεν θα πρέπει να εργάζεται ε, με όρους επισφαλούς και αναξιοπρεπούς εργασίας όπως είναι η μαύρη εργασία, η παράνομη και η ε, ε, ψευδός αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν. Πολλές φορές είναι και παράνομοι οι εργαζόμενοι αυτοί. αλλά ε, θα πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι καταστάσεις και να ε, περιοριστούν πριν ε, κυριαρχήσει μια γενική υποψία για όλο τον κλάδο. Ευχαριστώ κύριε Κρότσμαν, κυρία Ρούλε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έχει κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν έχουμε προβλήματα με τις προτάσεις του. Μια ερώτηση έχω εγώ προς τον κύριο Κρότσμαν. Έχει κάνει μια τροπολογία παριθμών 17 Μ' αρέσει αυτό για τους δείκτες ποιοτικού των υπηρεσιών, απλώς απορώ. Γιατί το κάνετε και θέλετε να συμμετέχουν μόνο οι εργοδότες και εργαζόμενοι χωρίς τα συνδικάτα. Πού το είδατε αυτό τα συνδικάτα. Όχι, όχι, εντάξει, ωραία την ευκαιρία να λύνονται έτσι πολλά προβλήματα ε, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουμε εμείς σε λεπτομέρειες. Γιατί έχει δίκιο ο κύριος Άριας Τσεβερία. Ε, όταν βάζουμε τόσο πολλές τροπολογίες για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τότε η έκθεση ολόκληρη πηγαίνει προς μια τελείω διαφορετική κατεύθυνση και παίρνει μια άλλη χρειά. Οπότε θα αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν ασχολείται η Επιτροπή Απασχόλησης με αυτό το θέμα, γιατί κανονικά είναι δική τη υπόθεση. Όχι να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δείκτες ε, να εκπονήσει ε, για το σύστημα αξιοπιστίας, αλλά να συμμετέχουν παρακαλώ εκεί και τα συνδικάτα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέλη έχουν το λόγο. Ζήτησε το λόγο η κυρία Γκέπχαρτ, κάποια άλλη. Αντώνιο για τις τροπολογίες σου, κάποιος άλλος. Λοιπόν, η κυρία Γκέπχαρτ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Όντως έχω κάνει πολλές τροπολογίες μαζί με τη συνάδελφο Όλγα Σενάλοβα που ε, έχουν να κάνουν ακριβώς με τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν αυτό το καιρό ε, και δεν είναι τίποτα ε, ανεδαφικές αιτιάσεις κύριε Κρόιτσμαντ και, και πράγματα που δεν ευσταθούν. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μας τα έχουν πει αυτά και οι εργαζόμενοι εκεί. Δεν είναι καθόλου βάσιμα λοιπόν. Ξέρουμε πώς δουλεύουν εκεί. Είναι τεράστια η πίεση του ανταγωνισμού σε πολλές εταιρείε και δεν δέχομαι αυτό να είναι εις βάρος ε, των εργαζομένων εκεί, ανδρών και γυναικών. Επίσης δεν θα πρέπει να λησμονούμε εδώ ότι εκτός από ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουμε ακόμα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα που θέλουν να επιβιώσουν. Και είναι θέμητος αυτός ο ανταγωνισμός, ε, ακριβώς λόγω αυτών των κακών συνθήκων εργασίας. Και δεν μπορούν να επιβιώσουν, θα βάλουν λουκέτο τα μαγαζιά αυτά, γιατί ακριβώς ε, είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν με σωστές συνθήκες και απασχόλησης και πληρώνουν κανονικά τους εργαζομένους τους. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Όλο αυτό το πλέγμα δεν επιτρέπεται να το λησμονίσουμε. Γι' αυτό κάναμε τις τροπολογίες έτσι ώστε να μην λησμονηθεί αυτή η διάσταση. Λοιπόν, η πρόταση, η τροπολογία 17 Ε, με την ε, προσθήκη της κυρίας Ρούλε θεωρώ ότι έχει νόημα, χωρίς να προεξοφλώ αυτά που θα πει Όλγα Σανάλοβα που είναι η σκιώδης μας εισηγήτρια, αλλά έτσι δεν αναιρούνται καμία περίπτωση οι δικές μας τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί αλλού. Ευχαριστώ. Ωραία. Όπως βλέπετε φωτίζονται οι εξελίξεις, ανεβαίνουν και οι και τα Ο Δεκάμπος. Ευχαριστώ Μάλκομ υπέβαλα προτάσεις τροποποίησης που είχαν στόχο να βελτιώσουν την έκθεση και που είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που έγιναν στην ομάδα εργασίας e-commerce όπου είχαμε μετάσχει. Χαίρομαι που βλέπω ότι η πλειοψηφία των τροπολογιών αυτών έγινε δεκτή και ότι υπάρχει και ότι υπάρχουν απόψεις που συγκλίνουν προ την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα για να μην ξεκινήσει ένα κοινωνικό dumping. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια σειρά ευκαιριών για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να λάβει κίνητρα για να μπορέσει να εμπνεύσει στους καταναλωτές εμπιστοσύνη. Και νομίζω η λέξη κλειδί είναι εμπιστοσύνη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια αγορά παραδόσεων με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα που προσαρμόζεται και στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή. Θεωρούμε σημαντικό επιπλέον η Επιτροπή να ενισχύσει τη δημιουργία ε, online ιστοσελίδων για να μπορεί να υπάρχουν συγκρίσεις των υπηρεσιών των διαφόρων εταιριών παραδόσεων σε πολλές γλώσσες ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορεί να λάβουν μία απόφαση με πλήρη επίγνωση και των τιμών και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Είμαι πεπισμένος ότι το κείμενο αυτό θα βελτιωθεί με την ε, συνεισφορά των συναδέλφων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητής, ιδίως δε, να ευχαριστήσω τον κύριο Άρης για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Ευχαριστώ. Ωραία. Κάποιος άλλος. Α, ξεχάσαμε την Επιτροπή, απλά πείτε μας ποιος είστε. Και με χαρά θα ακούσουμε τα σχόλιά σας για τις τοπολογίες Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σβάμπε, εξ ονόματος του εισηγητού. Ευχαριστώ. Είμαι επικεφαλής ε, της ε, ομάδας στην Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο σήμερα για την ε, πολύ καλή για τα πολύ καλά σχόλιά τους. Θα περιοριστώ σε μια σειρά παρατηρήσεων. Πρώτα πρώτα να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αναγγείλαμε ότι θα προχωρήσουμε με έναν οδικό χάρτη, πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση του περάσματος ε, στην ε, ενιαία αγορά παράδοσης δεμάτων. Ελπίζουμε το κολέγιο των επιτροπών θα μπορέσει να εγκρίνει τον οδικό χάρτη σύντομα, δηλαδή πριν τελειώσει το έτος. Ελπίζουμε λοιπόν τις επόμενες δύο εβδομάδες να λάβετε κι εσείς γνώση των δράσεων που έχουμε αναγγείλει στον οδικό χάρτη έγκαιρα για την χριστουγεννιάτικη περίοδο. Το τι θα περιλάβει τώρα ο Οδικός χάρτης. Οι στόχοι που συζητήθηκαν θα εμφανιστούν προφανώ στον οδικό χάρτη. Διαφάνεια και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η διαφάνεια είναι σημαντική και για του λιανέμπορου και για, τους, ε, και για τις ταχυδρομικέ υπηρεσίε και για του καταναλωτέ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, και αυτό αναφέρθηκε ήδη και σήμερα. Οπότε θα περιλάβουμε συγκεκριμένα συγκεκριμένα στοιχεία για υποχρεώσεων, για τις υποχρεώσεις παράδοσης του ηλεκτρονικού εμπόδιο. Ο δεύτερος στόχος θα είναι να ενισχύσουμε την διαθεσιμότητα λύσεων παράδοσης. Και αυτό είναι ένα θέμα που σχετίζεται με την σύνδεση της διαλειτουργικότητας, της ανάπτυξης ανοιχτού interface. Εν τέλει, αν υπάρχουν περισσότερες πλατφόρμες που προσφέρουν προϊόντα στην αγορά, θα έχουμε αυτόματα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και, για παράδειγμα, θα δώσει καλύτερη δυνατότητα χρήσης της ενοποίησης μικρών όγκων παράδοσης και λόγω της αυξανόμενης αποτελεσματικότητας ακριβώς, ελπίζουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του κοινωνικού ντάμπινγκ που αναφέρθηκε προηγουμένως. Όλοι συμφωνούμε και η Επιτροπή ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μείωση των συνθήκων εργασίας των ε, τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να γίνουν σεβαστές όπως έχουν συμφωνηθεί σε νομικό επίπεδο και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για, και για τα συνδικάτα βεβαίως. Τρίτον, Κύριος στόχος μας είναι η αύξηση του μηχανισμού αντιμετώπισης των καταγγελιών και του μηχανισμού αποκατάστασης ζημιών για τους καταναλωτές. Προφανώς αυτοί κινούν την αγορά και αυτό το θέμα θα το εξετάσουμε ιδιαίτερα. Αυτά είναι τα σχόλια εξ ονόματος Επιτροπής. Προφανώς, όπως ήδη αναφέρθηκε εισαγωγικά, δεν θα υποβάλουμε πρόταση ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμένου στη φάση αυτή. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Τέμινγκ, έχετε ξανά αφήσει συναντήσεις με συγγνώμη που δεν σας αναγνώρισα. Οι πληροφορίε που μας δώσετε για την δημοσιοποίηση ενό οδικού χάρτου θα είναι σημαντικέ για τον εισηγητή. Οπότε στην επόμενη συνάντηση 27-28 Νοεμβρίου που θα εξεταστούν οι συμβασικέ τροπολογίε, θα έλεγα το εξή: Αν έχει βγει ήδη ο οδικό χάρτη, θα ήταν μια ευκαιρία να συμπεριλάβουμε συμβασικές τοπολογίες που θα λάβουν υπόψη και τον οδικό χάρτη. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέλουμε ενημερωμένη έκθεση και, και κάπως θα πρέπει να το χειριστούμε το θέμα του οδικού χάρτη. Πάντως αρμοδιότητα του εισηγητή είναι. Ο στόχος ήταν να ψηφιστεί 27-28 και να περάσει τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια. Δεν είναι όμως νομοθετικό κείμενο. Υπάρχει λοιπόν μια ευελιξία. Αν θέλει και ο εισηγητής να δει και τον οδικό χάρτη να το δούμε. Τέλος πάντων, ο κύριο Φάμπε θέλει να παρουσιάσει κάποιες σκέψεις εξ όνομα του κύριου Αρίας. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Να σας ε, ενημερώσω ότι θέλουμε να ξέρουμε κάθε εξέλιξη από πλευρά Επιτροπή στο συντομότερο δυνατό για να μπορέσουμε να κάνουμε την έκθεση αυτή όσο πιο ενημερωμένη γίνεται. Θα περάσω τα μηνύματα όλων των συναδέλφων στον ε, συνάδελφο κύριο Αρίας και όταν επιστρέψει από την Ισπανία είμαι βέβαιος ότι θα έχει και ενέργεια και βούληση να αντιμετωπίσει με συμβιβαστικό και αποτελεσματικό τρόπο τα κείμενα. Η σημασία είναι να σταθούμε στα βασικά του ζητήματος, όχι να λάβουμε υπόψη ό,τι προκύψει. Έρχονται και τα Χριστούγεννα, οπότε όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 10 παρατέτω θα ξεκινούσαν οι εξελίξει, οι ψηφοφορίε. Ε, προλάβαμε και τελειώσαμε. Αν θέλετε, πηγαίνετε να πιείτε έναν καφέ, αλλά μην χαθείτε, γιατί θέλω να ξεκινήσω στι παρατέτω ακριβώ τι ψηφοφορίε. Γιατί μέχρι τις 11 το θα ψηφίζουμε. Διακοπή 10 λεπτών.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Uh, sorry a bit late, but we had one or two um, issues on the voting list for Mr. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα με την έκθεση De Jong. Θα τα πούμε αργότερα όμως αυτά. Καλώς ήρθατε στη ψηφοφορία μας για σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε πολλοί. Λοιπόν, θα υποφεληθώ να σας πω ότι ξέρω πολλοί συνάδελφοι συμμετείχαν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τον μήνα για την ενιαία αγορά. Ο κύριος Μπαρνιέ μου έστειλε μια επιστολή πολύ επενετική που λέει ότι 6.500 άτομα ε, παρακολούθησαν 84 ε, chat και 55 ηλεκτρονικές πλατφόρμες παρακολουθώντας 786 προτάσεις είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και θα ήθελα δημοσίως να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που δούλεψαν για την ιδέα του μήνα της ενιαίας αγοράς και όλοι συμμετείχαν, όσοι συμμετείχαν στις ε, live αυτές τις συζητήσεις στα chat. Βλέπω ότι κουνάει το κεφάλι της η κυρία Στάιλερ. Πάντως πήγαν πολύ καλά τα πράγματα και ο κύριος Μπαρνιέ το εκτίμησε όλο ιδιαίτερος. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες μας για σήμερα. Πρέπει να ψηφίσουμε για τις ε, διαπραγματευτικές εντολές για πολλά ζητήματα και πρέπει επίσης επισήμως να εγκρίνουμε τις, τα συμπεράσματα ε, των συνδιαλλαγών για κάποια θέματα. Έχουμε τα θέματα τη ασφάλεια αγοράς και τη εποπτεία αγοράς που θα τα πάρουμε ως πακέτο και γι' αυτό προτείνω να τα, τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Κυρία κάνουν δεν εδώ, αλλά τέλος πάντων μου φαίνεται λογικό αυτό. Να πω επίσης ότι η διαπραγματευτική εντολή συζητήθηκε εκτενώς από τους συντονιστές και ξέρω ότι ε, υπήρξαν εξελίξεις. Ίσως ε, ο κύριος να, η κυρία Σαλντεμόζε να μπορεί να μας πει περισσότερα πράγματα για το πώς ε, έχει η κατάσταση. Για το κατά πόσο θα λάβουν την εντολή οι κυρίες Σάλτεμόζο και Πιετικάνεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι πιστεύω ότι χρειάζεται να ζητήσουμε εντολή διαπραγματευτική γιατί έχουμε ευρεία ε, συνένεση που να υποστηρίζει την έκθεση και νομίζω ότι είναι ε, δυνατό να υπάρξει αποτέλεσμα κατά τις διαπραγματεύσεις και το Συμβούλιο προτίθεται να εξέδει τις λύσεις, θα είναι καλό και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει είναι Κατά την ε, ψηφοφορία είχαμε αυτή την ε, πρόταση για την ασφάλεια της αγοράς και δεν ήταν τμήμα αυτό της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο να ζητήσουμε μια μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου από αυτού και συμφωνήσαμε με τους σκιώδεις εισηγητές ότι θα ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για τις συνέπειες. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες και για τις διαπραγματεύσεις μας. Επίσης θα συλλέξουμε πληροφορίες και για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα ε, τις απαιτήσει για τους οικονομικούς ε, φορείς, αλλά μόνο για το, ε, το σήμα ασφάλειας θα ζητήσουμε την εντολή. Πρέπει να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και ούτως ή άλλως θα ενημερώνουμε την Επιτροπή για τις εξελίξεις. Ελπίζουμε ότι θα μας υποστηρίξετε. Υπάρχει ευρεία συνένεση πίσω από την έκθεση, γι' αυτό ζητούμε την εντολή αυτή. Πρόεδρος. Ούτω ή άλλω έχουμε δρομολογήσει πολλέ μελέτε ε, για την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων αυτών, κύριο Κρόιτσμαν. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με τι διαπραγματεύσει, αλλά. Όσον αφορά τη μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου, ο κύριος Φαμπ είχε ζητήσει μία ξεχωριστή για το σήμα ασφάλειας και για το Made in. Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μεγάλο το πρόβλημα της ε, ε, ε Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η τεράστια αξιολόγηση αντικτύπου για να ξέρουμε τι αντίκτυπος θα υπάρχει και ε, στα δύο θέματα. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Ούτως ή άλλως ε, προγραμματίζουμε ε, για το σήμα ασφάλειας ε, αξιολόγηση αντικτύπου, γιατί πιστεύει η κυρία Σαλντεμόζη ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε πραγματεύσεις όσον αφορά το σήμα προέλευσης. Σκοπό έχουμε να κάνουμε μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου για να αναλύσουμε την ίδια την ε, προοπτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και να δούμε και τον αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, θα ενημερώσουμε βέβαια του και τους συζητητές τους ή άλλως αυτό το τμήμα της ενημέρωσης. Δεν υπάρχει λόγος, αφού θα κάνουμε και εμείς, να κάνουμε και εμείς ε, αξιολόγηση αντικτύπου όταν έχει κάνει ήδη η αλλω αυτο το τμημα τη ενημέρωση. δεν υπαρχει λόγο, αφου θα κανουμε και εμει Επιτροπή. Υπάρχουν κάποια συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία έχουν αποσταλεί στου κοιόδη Αλλά όσον αφορά τη διαπραγματευτική ομάδα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ του. Αν χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, μπορώ τότε να σα ζητήσω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώ. Να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά ή αποχή σε σχέση με το κατά πόσο θα λάβει η διαπραγματευτική ομάδα εντολή. Άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία Πέντρικαστ δεν έχει την κάρτα της. Πέρας ψηφοφορίας. 33-33. 33-0, ε, συγγνώμη. 34. Έχετε την ε, διαπραγματευτική εντολή λοιπόν. Συγχαρητήρια. Τώρα να επιβεβαιώσουμε τη διαπραγματευτική θέση. Α, ο κύριος Ροσφόρ πρώτα και μετά η κυρία Ρόιτοβα. Α, πρώτα η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι δεν μπόρεσα να ψηφίσω γιατί έχει πρόβλημα το μηχάνημά μου. Ναι, θα δούμε. Θα βεβαιωθούμε ότι δουλεύει καλά η κάρτα σας. Λοιπόν, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων τριμερούς διαλόγου. Χθε, ο κύριος Ροσφόρ μας είπε για την έκβαση του προγράμματος για τους καταναλωτές 2014 2020. Δεν είναι εδώ όμως σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα, ο συμβασμός με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λέω για όσου δεν ήταν εδώ χθε. Τώρα προσπαθούμε να δούμε τον προπολογισμό του προγράμματος. Εκ μέρου του κ. Ροσφόρ και ως πρόεδρος της διαπραγματευτική ομάδας θα ήθελα να σας καλέσω να εγκρίνετε, να εγκρίνουμε τις τελικές λεπτομέρειες έκθεσης. Το σημαντικό ήταν ε, έχουμε ένα δικαίωμα παρακολούθησης για τη χρήση των ε, ταμείων και την εφαρμογή των στόχων στο πρόγραμμα και όπως επίσης και για τη διαχείριση του προγράμματος. Θα υπάρξει μια πλήρης μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση για να ελέγξουμε την πρόοδο των διαφόρων προγραμμάτων και να ε, κάνουμε προσαρμογές αν χρειαστεί. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία. Αν δεν θέλει κανείς από τους σκιώδεις να λάβει το λόγο, να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ηλεκτρονικός και πάλι για την επίσημη έγκριση του προγράμματος καταναλωτών, το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής. Η κυρία Πέντεγκαστ ψηφίζει υπέρ. Η κυρία Ροϊτόβα εξακολουθεί να έχει πρόβλημα. Α, όχι, εντάξει, δουλεύει τώρα η κάρτα. Πέρα της ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές. 32 και 2 αποχές. Πάμε λοιπόν τώρα στο πακέτο Ρόιτοβα. Λέω να τα ψηφίσουμε όλα μαζί αυτά τα θέματα ευθυγράμμισης και αναδιατύπωσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διατήρηση των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ομάδες εργασίας και άλλες πτυχές των διαπραγματεύσεων. Κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρίως για τη βοήθεια, τη μεγάλη υπομονή σας και την προθυμία όλων των σκιωδών και της γραμματείας και ε, του Προεδρείου της Επιτροπής. Ήταν πολύ μακρά η διαδικασία αυτή. Ε, πετύχαμε πάρα πολλά. Δεν ήταν μόνο επί της ουσίας. Ε, γενικότερα έγινε μεγάλη συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου ακριβώς ε, για το ρόλο πρώτα του Συμβουλίου και μετά του Κοινοβουλίου και πώς θα συμμετέχει ε, στις λεγόμενες διαδικασίες της επιτροπολογίας. Και καταλήξαμε σε μια συμφωνία ε, που μας επιτρέπει σήμερα να ψηφίσουμε όλη αυτή τη δέσμη. Στην Ολομέλεια θα αναγνώσω μια δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα και βάσει όλων αυτών βασιζόμαστε και ισχύει ε, το άρθρο 15 της Διοργανικής Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ορίζουμε σαφώς και διαπαντός ε, τα διαδικαστικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, αυτό είναι θέμα βεβαίω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά όταν υπάρχουν επιτροπές εμπειρογνωμόνων και ασχολούνται με άλλα θέματα εκτός του αντικειμένου τους, πρέπει να έχουν διαφορετική σύνθεση και στη σύνθεση αυτή πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λαμβάνει όλα τα έγγραφα και όλη την ε, ενημέρωση. Αυτό είναι το κλειδί της ε, διαμάχης που είχαμε και το διαπληκτισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα που δίρκησε 18 μήνες. Δυστυχώς τώρα θα πρέπει να περιμένουμε και τη γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής και μάλλον θα χρειαστεί χωριστή ψηφοφορία. Αυτά και σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε ε, πλέον στην ε, ολοκλήρωση αυτής της μακράς διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much for leading that. Ευχαριστώ. Επίσημα το θέτω να επιβεβαιώσω ότι επήλθε συμφωνία για μια αιτιολογική σχέση μετά από πολλές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Εν μέρει ωστόσο η συμφωνία περιλαμβάνει ότι πρέπει να υπάρξει επίσημη δήλωση του Κοινοβουλίου που θα παρατηθεί στο επίσημο, σε μια σειρά ε, φίλων της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα σας τα διαβάσει περισσότερο η Σουζάνα. Το κείμενο λέει «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο μόνο και στο μέτρο των εφαρμοστικών πράξεων βάσει του κανονισμού 182 του 2011 θα συζητούνται σε συναντήσεις επιτροπών και μόνο τότε μπορεί τούτο να θεωρηθούν ε, ως επιτροπές επιτροπολογίες βάσει του παρατήματος 1 της Συμφωνίας Πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών που υπάγονται κατά βάση, ε, ως, ως εκ τούτο στο σημείο 15 της Συμφωνίας Πλαίσιο όταν άλλα θέματα συμφωνούνται, συζητούνται, δεν θεωρούνται ε, επιτροπές επιτροπολογίας. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο, αλλά εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας να μετέχουμε σε συναντήσεις που αφορούν θέματα εκτός του πεδίου εφαρμογής των εφαρμοστικών πράξεων, των εκτελεστικών πράξεων και ε, δεν ήταν σαφές στη συνάντηση. Κάποια κράτη-μέλη αμφισβήτησαν την δυνατότητα αυτή, προσπαθήσαμε να τους πείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εμένουμε λοιπόν στη διαφύλαξη των ε, αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Προτείνουμε λοιπόν το πακέτο με την συγκεκριμένη δήλωση ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας σοσιαλιστής παραπάνω. That's fine. Okay. Yep. Okay. Mm. <laughs> uh, Right, the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 33, 33 υπέρ, ουδής κατά. Ευχαριστώ τη Σουζάνα που ήταν πολύ υπομονητική για τη διάρκεια των μακρών διαπραγματεύσεων. Προχωρούμε. Άλλες ψηφοφορίες. γνωμοδότηση Κόρατσα Μπίλτς για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επιστημιστική κρίση, περιπτώσει απάντηση στην τροφική αλυσίδα και καταπολέμηση αυτών των πρακτικών. Άννα, κάτι? Να ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ελπίζω να ικανοποιηθούν όλοι, να είναι ικανοποιημένοι όλοι με, τη συμβαστική, με το συμβαστικό κείμενο που επιτύχαμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Και αυτό απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Ηλεκτρονικά θα γίνει για να γίνει ο έλεγχος. Για τη συμβαστική 1 λοιπόν. Πάλι ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 17 με 15. Άρα οι 3 και οι 5 καταπίπτουν. απολογία 4 υπέρ. Κατά. Απολύπτεται. 7 υπέρ. Sorry, I had the wrong voting list, apparently. Συγγνώμη, από ό,τι φαίνεται έχω λάθος κατάλογο ψηφοφοριών. Κατά τμήματα ψηφίζουμε την τροπολογία 7. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 7 υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γι' αυτό. Για το πρώτο τμήμα της 7. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 5 υπέρ 18 κατά. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. 6. Με μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Με την προφορική τροπολογία. 8 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 11 σαν προσθήκη. Υπέρ κατά και αυτή δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή 29 υπέρ 2 κατά 2 εποχές. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Κορατσαμπίλτ. Περιμένουμε να υποστηρίξετε την απόψή μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προχωρούμε τώρα. Έκθεση Μπάστος για την Νομική Επιτροπή. Δύο εκθέσεις. Για τον κανονισμό σχετικά με το κοινοτικό σήμα Το πρώτο όμως που ψηφίζουμε είναι για την οδηγία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα σήματα. Το έχετε? Άρθρο 3. Παράγραφος 1. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 σαν προσθήκη, ως προσθήκη υπέρ, κατά, δεκτή. 5 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 6 μπάστος, υπέρ, κατά, δεκτή. Τι ψηφίζουμε πρόεδρε, την οδηγία ή τον κανονισμό. Την οδηγία είπα, λέει ο πρόεδρος. on... Uh, did you want to start again? Sorry. No. Θέλετε να ξαναρχίσουμε. Όχι. Μπερδεύτηκα. Όταν αναφέρετε ότι θα ψηφίσουμε την τροπολογία 9. Δεν έχω 9 εγώ στο δικό μου κατάλογο. Mm. I didn't think I said nine, actually. I didn't say nine, I said six. Δεν είπα εννέα, έξι είπα. I said six, I think. All right, sorry, this is slightly confusing because we have two. Συγγνώμη, υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα λόγω του ότι υπάρχουν δύο γνωμοδοτήσει μπάστους. Η σύντομη θα γίνει πρώτα, δηλαδή η οδηγία για την προσέγγιση της νομοθεσία σχετικά με τον σχετικά με το κοινωνικό με το σήμα, αναδιατύπωση. Συμφωνείτε όλοι. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε. Τέσσερα μπάστος για το άρθρο 3 παράγραφος 1 β. Λοιπόν, ξεπερνάμε τα πρώτα. Τέσσερα υπέρ. Κατά δεκτή. 17 ως προσθήκη υπέρ, κατά, δεκτή. 5 υπέρ, κατά, δεκτή. 6 υπέρ, κατά, δεκτή. 18 παντζέρι υπέρ, κατά, δεκτή. 19 έγκστρομ υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 20 κατά τμήματα, κύριε Μπάστος. η ομάδα είναι κατά, η ομάδα μου είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας. Θέλουμε να ψηφιστεί το υπόλοιπο τμήμα χωρίς την προφορική τροπολογία. Την αρχική τροπολογία δηλαδή. Τι είναι, μια προσθήκη δύο λέξεων, and distribution. Μια ομάδα είναι κατά. Πρόεδρε, να κάνω ένα σχόλιο. Αν κατάλαβα καλά, δεν είναι αντίθετη με το περιεχόμενο της τροπολογίας, αλλά για διαδικαστικούς λόγους, επειδή είναι συμβαστικό κείμενο, πρέπει να είμαστε κατά. Είχα μια ανταλλαγή απόψε με τους φιλελεύθερους που δεν κατάλαβαν γιατί ήμασταν κατά. Εμείς θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε, αλλά ο σύμβουλος μου είπε ότι πρέπει να αρνηθούμε αυτή την προφορική τροπολογία. Μα δεν είναι συμβαστική τροπολογία, μια τροπολογία είναι. Ζητείτε κατά τμήματα ψηφοφορία στην τροπολογία 20, δεν είναι συμβαστική. Ο κύριος Κρόιτσμαν πρότεινε μια προφορική τροπολογία που δεν θέλει συγκίτρια, αν κατάλαβα καλά. Στο πρώτο τμήμα. Και στο δεύτερο τμήμα υπάρχουν προφορικές τροπολογίες. Πρόεδρε, το ΕΛΚ είναι κατά της προφορικής τροπολογίας Και με τον τρόπο αυτό ψηφίζεται η τροπολογία του ΕΛΚΑ που ήταν η αρχική τροπολογία. Είναι απλό, πρόεδρε. Δηλαδή δεν λαμβάνουμε υπόψη την προφορική τροπολογία. Αυτή είναι η θέση μας. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Το αρχικό κείμενο της τροπολογίας. κατά δεκτή. Δεύτερο τμήμα, όπως είναι κατατεθειμένο εδώ, χωρίς προφορική τοπολογία, δεν έχει δηλαδή, υπέρ του δεύτερου τμήματος. So we need to vote the second part. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Οι υπογραμμισμένε λέξει είναι η τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. 21. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 23. στο, στην, στον κατάλογο βλέπετε ότι ένα τμήμα της τροπολογίας έχει αποσυρθεί. Η 23 όπως άλλαξε, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά θα το κάνουμε. Γιατί τσίμα τσίμα το βλέπω. 23. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτό. 18-14. Η 7 Μπάστος υπέρ κατά ως προσθήκη δεκτή γίνεται ως προσθήκη όμως είναι, είναι σαφές 22 πάλι ως προσθήκη υπέρ κατά δεκτή 24 υπέρ κατά απορρίπτεται 25 υπέρ κατά δεκτή 26 υπέρ κατά απορρίπτεται. 8 συγγνώμη κύριε Μάγερ. υπέρ κατά δεκτή. 9 υπέρ κατά δεκτή. 27 και 28 καταπίπτουν. 29 υπέρ κατά δεκτή. 30 υπέρ κατά δεκτή. 31 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 32. Αποσύρθηκε η τελευταία φράση. Ποιο είναι, ποιοι είναι υπέρ της 32 χωρίς αυτό. Δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Έλεγχος της 33. Ψηφίζουμε. στις πληροφορίες. Απορρίπτεται. 17 για την κύριε και κύριε Πρίντο για την εκατά. 34 υπέρ κατά Και εδώ χρειάζεται έλεγχος. Ψηφίζουμε για την 34. Who is that? we got someone additional? Agustin Dras de Mera has been communicated. Yeah. He is voting for the Right, okay. The vote's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Και αυτή απορρίπτεται. Πάλι με μία ψήφο. Το 35. Υπέρ. Και εδώ ψηφίζουμε πάλι ηλεκτρονικά γιατί όλα τσίμα τσίμα βγαίνουν. 33 πρέπει να είναι τα άτομα που ψηφίζουν. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 16 προς 14. Και δύο εποχές. Καταπίπτει 36. Αιτιολογικές σκέψεις. Οι 10 και 11 εγκρίθηκαν αυτόματα. Οι 12 που είναι οι μόνοι υποψηφισμοί, γιατί όλες οι άλλες ε, είναι, γίνονται δεκτές αυτόματα, χωρίς ψηφοφορία. 12 υπέρ κατά δεκτή. Άρα αν κατάλαβα καλά κύριε Μπάστος, εγκρίνονται αυτόματα όλες οι άλλες αιτιολογικές σκέψει. Πάμε στην τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε για την γνωμοδότηση Μπάστο. Βιαστείτε. «32 υπέρ, καμία ψήφος κατά μία αποχή. Ευχαριστούμε κύριε Μπάστος. Προχωρούμε. Δεύτερη έκθεση Μπάστος. πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα πάλι. Τοπολογία 4, υπέρ. Κατά, δεκτή. 23, υπέρ. Κατά, δεκτή. 24, υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. Και εδώ πάλι είστε κατά της προφορικής τροπολογίας γιατί είναι το ίδιο κείμενο. Ναι. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 25 χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχαιρετή δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεκτή. 26 υπέρ κατά απορρίπτεται. 27 όπως με τις αλλαγές που έχουμε υπέρ, κατά. υπέρ Θέλετε να ψηφίσουμε. 27. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, 14 κατά. 15-15. Καταπίπτει. Η κυρία Πρέντεγκαρντ είναι κατά. Θα uh, ήταν... Uh, Ψηφίστε, And then we κύριε Βερνιό, καλύτερα να ψηφίσει κύριε Βερνιό παρά εσείς αν δεν σας πειράζει. Νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Θα ψηφίσει η κυρία Βερνιό με τους ε, σοσιαλιστές. Επαναλαμβάνει την ψηφοφορία. αυτό υπάρχει ένας έξτρα βουλευτής από το ΕΛΚ. Is he still within the numbers? Yes, he is. You sure? Yes, they have double checked. We have Mr. Diaz de Mera, who is voting with the EPP. Η κυρία Diaz de Mera ψηφίζει με το ΕΛΚ χωρίς... Ο κύριος χωρίς κάρτα. Ψηφίζω με το ΕΛΚ, δεν έχω κάρτα, να λαμβάνετε υπόψη ότι θα σηκώνω το χέρι μου όποτε ψηφίζω. Δεν μπορείτε να στείλετε κάποιον να σας φέρει την κάρτα σας και διέστε μέρα. Σπίτι μου είναι η κάρτα, οπότε θα αργήσει κάπως. Δεν μπορούν να σας βγάλουν διπλή κάρτα οι υπηρεσίες μας. Στείλτε κάποιον ε, στο γραφείο από κάτω να σας βγάλουν δεύτερη κάρτα. Εντάξει πρόεδρε. 34 είμαστε ψηφίζ... Πάλι 16-16 είναι. Όχι, δε... Δε... κερδίζει γιατί ο κύριος Δίας Δεμέρα ψηφίζει προφορικά. Οι falls. Η, η καταπίπτει πάντως. 28 Κρόιτσμαν. Προχωράμε. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 29 Παντσέρι. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 30. Προσπαθούσα να προχωρήσω πολύ γρήγορα η τροπολογία 5 της εισηγήτριας μπορεί να ως, να ψηφιστεί ως προσφύκη στην 26. Άρα την 5 ψηφίζουμε τώρα. Δεν την ψηφίσαμε. Εγώ νόμισα. Δεν διάβασα ό,τι όλες. Δεν καταπίπτει. Ως προσφύκη μπορεί να ψηφιστεί. Δεν διάβασα καλά τον κατάλογό μου, κύριε Γκέπχαρτ. Η πέντε, ως προσφύκη, υπέρ, κατά, δεκτή. Ξαναπάμε τώρα στην 30. Η οποία καταπίπτει όμως, γιατί εγκρίναμε την 29. 31. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή και η 7 ως προσφύκη υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 Κρόιτσμαν υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 καταπίπτη, 36 υπέρ υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά δεκτή 38 υπέρ κατά δεκτή 39 και 40 μαζί υπέρ, κατά, δεκτές. 9 υπέρ, κατά, δεκτή. 11 υπέρ, κατά, δεκτή. 12. Τη 10 δεν ψηφίσαμε υπέρ. 10, 11, 12 μαζί. Οι τρεις τροπολογίες 10, 11, 12. Στην ίδια παραγραφή είναι όλες. Υπέρ των τριών κατά δεκτές 41 συγγνώμη υπέρ κατά απολύπτεται Τώρα θα κάνουμε έναν έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία για τη 41 ο κ. Δίας Δεμέρα είναι υπέρ πέρας ψηφοφορίας δεκτή 42 υπέρ. Δεκτή. 13 υπέρ. Δεκτή. 43. Εγκρίθηκε με την 42. Ε, 45 υπέρ. Κατά. Δεκτή. πίπτη 44. 47 υπέρ. Κατά. Δεκτές καταπίπτει 46. 48 και 49 μαζί, υπέρ, κατά. 50 δεν ψηφίζεται, 14 υπέρ, κατά, δεκτή 51 πίπτη. Αιτιολογικές σκέψεις, 15 υπέρ, κατά, δεκτή, 16 υπέρ, κατά, Αποχές δεκτή. 17, 18, 19 εγκρίνονται αυτό μετά 20 υπέρ κατά δεκτή και 22 υπέρ κατά δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 34 υπέρ, μία κατά καμία αποχή. 35 στην πραγματικότητα γιατί είναι και ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστούμε την κυρία Μπάστος. Περιμένουμε να υποστήριξετε τη θέση μας στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Προχωρούμε στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράση για το Γενικό Εμπόριο Πεσοφερσών των Παραγόντων. Ο κύριος Ντεγιόγκ είναι ο εισηγητή. Θέλει να πει κάτι, Κορνέλης. Πολύ σύντομα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω βεβαίω όλου και οδησίτες που μέχρι χτε εργάστηκαν σκληρά και μέχρι τη νύχτα για να επιτευχθεί όσο γίνεται μεγαλύτερο συμβιβασμό. Όταν φτάσουμε στην παράγραφο 9 θα ήθελα να επανέλθω για τον κατάλογο ψηφοφορία που δεν συνάδει ακριβώ με τι τελευταίε εξελίξει. Ευχαριστώ. Okay. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στην παραγραφωνία θα το δούμε, αλλά νομίζω ότι ήδη έχει προαναγγελθεί αυτή η αλλαγή. Απλώ θέλω να εξασφαλίσω να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο ότι έχουμε όλοι το σωστό κατάλογο μπροστά μας. Τον ίδιο κατάλογο. Λοιπόν, αρχίσουμε. Τροπολογία 13. Πέρες, υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να κάνουμε έλεγχο. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ 19 κατά. Η, επιτροπή τροπολογίας, η τροπολογία της Επιτροπής Διπλώμη καλύπτεται. Οπότε πάμε στην 3, κατά τμήματα ψηφοφορία. Έχει ζητηθεί από το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα τη συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα λοιπόν. Τη συμβαστική τροπολογία 3. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 16 κατά. Α, ο κύριος Δίας Δεμέρα έχει κάρτα. Έχετε μία ακόμη κάρτα. Μπράβο, δίκιο είχα. Λοιπόν, μέχρι και η κυρία Πέντεκαστ μπορεί να έχει κάρτα. Λοιπόν, έμπλεο, 19, 18 δεν την ψηφίζουμε, 19 στάιλερ, υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4α υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Οπότε τώρα Πάμε στην 23 ως προσθήκη. Που προστίθεται στη συμβιβαστική 4, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 26. Λόκεγκαρντ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογίε απασχόληση δεν τι ψηφίζουμε γιατί καλύπτονται. Πάμε στην 31 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Α, κατά τμήματα. <clears throat> Σωστά. Το ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής τροπολογίας 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Ως προσθήκη στη συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος πώς ψήφισαν οι φιλελεύθεροι, οπότε καλύτερα να την ελέγξουμε ηλεκτρονικό στη 40. 36 κάρτες βλέπω. Απορρίπτεται. 16-19. Λοιπόν, πάμε στη συμβιβαστική 8, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω τώρα έχουμε αλλαγή. Ντένις, θα ήθελες να μας πει ορισμένα πράγματα. Ναι, θα πρέπει να εξηγήσω. Εχθές προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για να συμπεριλάβουμε τι συμβιβαστικές 14 και τι τροπολογίες 44 και 45, αλλά δεν τα καταφέραμε. Χθε το βράδυ φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτό το κείμενο αυτό. Οπότε θα ήθελα να διατηρήσω στην παράγραφο 9 μόνο το πρώτο τμήμα όπως ε, προτείνει, προτείνει η φιλελεύθερη στην τροπολογία 44 να γνωρίζει το δικαίωμα των τοπικών αρχών 40, 45 τα δικαιώματα όταν αυτό θα έχει αντίκτυπο ε, περιβαλλοντικό ή οικονομικό και τη 44 να την ψηφίσουμε σαν προσθήκη, γιατί είναι συμβατές οι 44 και οι 45, απλώς η 44 προσθέτει νέα στοιχεία. Συμφωνείτε? Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική 14, όπως τη διάβασε ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη 44 ως προσθήκη στη συμβιβαστική υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Όχι, αυτή δεν είναι συμβιβαστική, είναι η τροπολογία 44. Η κυρία Κοράτσα Βίλτ λέει ότι υπάρχει αρνητικό πρόσημο στο κατάλογο. Πέρασε όμως η 14 συμβιβαστική, λέει ο πρόεδρος. Τώρα ψηφίζουμε τη 44 ως προσθήκη. Κυρία Κορατσαμπίλτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ. Κρίμα που τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία αλλάζει αυτό. Εγώ δεν θέλω το ΕΛΚ να πάρει την ευθύνη για το ότι δεν ψήφισε σωστά για τη συμβιβαστική 14. Θα ήθελα να σας ζητήσω ηλεκτρονικώς να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 14, αν δεν σας πειράζει. Συμφωνείτε όλοι, ο Εκτό μικροφώνου ο πρόεδρος, Δυστυχώ. Λοιπόν, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη συμβιβαστική 14. 35 κάρτες βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, πέρας ψηφοφορία, απορρίπτεται. Οπότε, συμβαστική τροπολογία 14 απορρίπτεται. Άρα τότε ψηφίζουμε ούτως ή άλλως 44. Όχι. Ναι, τη 44. Ψηφίζουμε τη 44. Ψηφίζουμε τη 44. Υπέρ. Όχι, καλύτερα ηλεκτρονικός διορθώνει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός τη 44. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα Στη 45 και 46. Α, καταπίπτουν αν, ψηφιστεί, αν υπερψηφιστεί 44. Οπότε πάμε στη 47, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 49, που είναι ε, συμβατή με τη 48, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50, υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό στην τροπολογία 50. Πέρας. All right. Are you sure? It's the Εγκρίνεται 18-16. Λοιπόν, 51. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 53. Με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Υπέρ κατά, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 22 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 55 με, με προφορική τροπολογία, όπως αναφέρεται στον κατάλογο, από την κυρία Κοράτσα Μπίλτ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 56 του εισηγητή, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. τρία της Επιτροπής Απασχόλησης. Είναι υπέρ της ε, τροπολογίας απασχόλησης υπαριθμών 2. Οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς ε, την τροπολογία αυτή, γιατί εγώ δεν κατάλαβα καθόλου ποιο ήταν το αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Παρακαλώ, οι συντονιστές να δείχνουν κυρίως των ε, φιλελευθέρων τι θέλουν να ψηφίσει η ομάδα τους πιο σύντομα ή δεν ξέρω να αποφασίζετε βλέποντας και κάνοντας ψηφίζετε. Λοιπόν, η κυρία Πρέντεργκαστ έχει επιτέλους κάρτα, τέλεια. Λοιπόν, 18 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται η κυρια πρεντεργκα εχει επιτελους καρτα τελεια λοιπον 18 υπερ 16 κατα εγκρινεται η τροπολογια 2 της απασχόλησης, 3 της απασχόλησης, υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Τώρα όλοι έχουν κάρτε. Mm. Κάποιος έχει κάρτα και δεν τη χρησιμοποιεί μάλιστα. Τέλο πάντων, πέρας πληροφορίε, απορρίπτεται αυτή η τροπολογία. Πάμε στη 12 με προφορική τροπολογία τη κυρία Κοράτσα Μπιλτ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 τη επιτροπή Απασχόληση. υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58 συμβατή με την 57 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15 της απασχόλησης με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κατά. Κύριε Μάτε ψηφίζετε. Α, ευχαριστώ πολύ. Κατά λοιπόν, σηκώστε τα χεράκια παρακαλώ. Το έλκει φωνή. Μα δεν ψηφίζει κανείς. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θα ήταν χρήσιμο να ψηφίζετε πάντως, να σηκώνετε τα χεράκια. Για την 58 μιλάω, που είναι συμβατή με την 57. Α, όχι, είμαστε στην Επιτροπή Απασχόλησης τώρα, τη 15 της Απασχόλησης. Διορθώνει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 59. ριγοιεν Πέρες. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5 της απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. έξι τη Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 7 τη επιτροπή απασχόληση με κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας αυτής. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει υποθέτω. Α, όχι, δεν καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 8 τη απασχόληση υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 11 τη επιτροπή απασχόληση υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 16 τη επιτροπή απασχόληση υπέρ, κατά, απορρίπτεται 19 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά απορρίπτεται 60 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική τροπολογία 9 πρώτο τμήμα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 17 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ, επαναλαμβάνω, κατά, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 65 ως προσθήκη υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 66. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Κατά τμήματα. Πρώτο. Τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 11. Το ΕΛΚ είναι υπεράριθμο κατά έναν. Κάποιος να μην ψηφίσει παρακαλώ. Από το ΕΛΚ. Εντάξει. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μία ψήφος διαφορά. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 73 καταπίπτει. 74 κατά πέπτη, 75 αποσύρθηκε, συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. Πάμε τώρα στην 83 για διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. να ψηφίσουμε την 83 ηλεκτρονικός, γιατί είναι σημαντική αυτή η τροπολογία και θέλω να είμαι βέβαιος. Έναρξη ψηφοφορίας λοιπόν για την 83. Πέρασε. Εγκρίνεται. 22-13. Άρα συμβαστική 13 καταπίπτει. Σε αυτή την περίπτωση Πάμε στην παράγραφο 20 τώρα. Τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός, Για την 89 μιλάω. Είναι πολλές οι ψήφοι κατά από ό,τι βλέπω. Άρα ψηφίζουμε την 89 ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Ευτυχώ το ελέγξαμε. 90 πίπτη. 91 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα σε αιτιολογικέ σκέψεις. Ένα και δύο μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, αιτιολογικές αναφορές. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά η φιλελεύθερη ψηφίζεται. Είστε εδώ. Ξανά. Τροπολογία 5. Υπέρ. Ποιος ψηφίζει υπέρ παρακαλώ. Για την 6, για την 6 διορθώνει ο πρόεδρο. 6, υπέρ. Συγγνώμη, μπερδευτικά. Το έχω μπερδεύσει τη γλώσσα μου. Λοιπόν, 6, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, ξύπνησαν και οι φιλελεύθεροι. 7. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Για την επτά μιλάω. Γεια σας κυρία Αντζελίλη. Καλώς ήρθατε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι ε, 11 και οι 12 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Α, όχι ξεχωριστά. Λοιπόν, 11 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 12 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου έκθεσης έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ, καμία ψηφο, κατά, αλλά 11 αποχέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντεγιόνγκ. Μήπω Μήπως θέλετε να μα πείτε τίποτα κύριε Ισηγητά. Πολύ σύντομα γιατί έχουμε και άλλε ψηφοφορίε και πάλι. Πιστεύω ε, ε, πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιοδησηγητές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους ανεξαρτήτους διανεμπόρους και για την καταπολέμηση των αθεμίτων εμπορικών πρακτικών. Έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την καθοδήγησή σας και χαίρομαι που συγκέντρωσε τόσο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Προχωρούμε λοιπόν και ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότης του κυρίου Μάγερ. Ε, θυμάστε για τα δικαιώματα των επιβατών ε, των αεροπορικών ε, εταιριών. Χάντς Πέτερ, θες να πεις τίποτα. Πολύ σύντομα, εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες και ιδιαίτερα ε, για αυτή τη σημαντική έκθεση. Είχαμε εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες email. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους και συγητές, γιατί θα έχουμε πει πολλές <laughs> φορές μαζί και με τον καθήλυνα αρμόδιο εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών, τον κύριο Μπαχ, και στα σημαντικά θέματα καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς, αλλά και σε άλλα, ίσως επιμέρους. Ε, και κύριε Πρόεδρε μπορεί να ψηφίσουμε και αμπλόκ πολλές φορές. Ε, βέβαια, ορισμένε ψηφοφορίε πρέπει να τι κάνουμε χωριστά, γιατί οι συμβιβασμοί σημαίνουν αλλαγέ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά καταπληκτική αυτή η συνεργασία μα. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Let's start then with 200. Ε, πάμε λοιπόν στην τροπολογία 200. Ψηφίπε. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Unblock τι μπορούμε να ψηφίσουμε. 16, 17, 18 μαζί γίνεται. Όχι. Αρχίσαμε. Ποιος είπε όχι. Η Άλντε. Καλώ του φιλελεύθερου. 16 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ε, θα μπορούσαμε να είχαμε ψηφίσει και μπλοκ, εν πάση περιπτώσει. 116-117 μαζί. Ψηφί υπέρ. Κατά αποχέ. Η προφορική τροπολογία του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική παρθόνα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 123 λοιπόν αμέσως. Υπέρ, κατά, αποχές, 124 προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 125 υπέρ, κα, υπέρ λέω, υπέρ ακόμα, κατά τώρα, εγκρίνεται σαφέστατα. 126 υπέρ υπέρ Μα δεν ψηφίζεται. That's really, that's rejected. 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20, 20, 20, 21, 22 μαζί ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 τι κάνει αυτή πίπτη. 129 προσθήκη ε, ψήφι υπέρ. Αυτές οι λέξεις που έχετε εδώ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 Θέλετε ηλεκτρονική απολύθευση. Συμβιβαστική υπαριθμών 2 λοιπόν. Εντάξει. Ψηφίζουμε. Εγώ νόμιζα ότι είχε εγκριθεί σαφέστατο. Συμβιβαστική 2 εγκρίνεται. Πέρασε. Ορίστε, 29 υπέρ 6 κατά. Καλά. Θέλετε να βεβαιωθείτε έτσι για καλό και για κακό. Ναι, τώρα κατάλαβα. <laughs> uh, right. Amendments one... Λοιπόν, 134, 135 τεχνικές είναι. 136 είπε κατά απορρίπτεται. Η 26 ε, του εισηγητή είπε κατά εγκρίνεται. 27 είπε κατά εγκρίνεται. 138 είπε Κατά. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 160 καταπέπτει. Η προφορική του εισηγητού τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 και 140 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι 30 και 142 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31 και 141 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 143. 44 και 45 μαζί υπέρ. Α, όχι, καταπίπτουν. Καταπίπτουν. Ναι, καλύπτονται από το 32, συγγνώμη. 33, ε, 147 και 148, είπε. Κατά. Εγκρίνονται. Η 146 λοιπόν καταπίπτει. 34, 149, 150 είπε. Κατά. Απορρίπτεται αυτή. Όλες αυτές. 151 τώρα. check. 34, 149 Λοιπόν, έλεγχος καλά. Πώς κάνετε έτσι. 34, 141 και 150. Εγκρίνονται μάλλον και καταπίπτει η επόμενη, 151. 35 του εισηγητού, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 152 καταπιπτεί 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 158 ως προσθήκη όμως. Υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 161, 2 μέχρι και 5 υπέρ. Είναι ταυτόσιμες. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 39, 166 μαζί υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 40 και 167 υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 168 και 69 μαζί, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 170 είπε. Κατά. Απορρίπτεται. Η 41 είπε. Κατά. Εγκρίνεται. 171 λοιπόν καταπίπτει. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. 173 και 174 δεν ψηφίζονται λέει. Α, ψηφίζω. Όχι. Όχι, δεν τις ψηφίζουμε. Πάμε στις 42. Ναι. Γιατί έχουν καλυφθεί. Έχουν εγκριθεί 168-69. Λοιπόν, 42 υπέρ. 42 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. is an addition to 170 or 241. 41, was adopted. It can be voted as an addition. Uh, now hold on, hold on. Μια στιγμή κάτι ελέγχουμε γιατί είναι λίγο μπέρδεμα εδώ. Σύμφωνα με τις συμβουλές που μας έχουν δώσει η 171 θα μπορούσε να ψηφίσει αυτή ως προσθήκη της 41 που εγκρίθηκε. Τι λέει ο συγητής. Συμφωνεί. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε την 171. Ως προσθήκη πάντα. 171 λέμε. Του κυρίου Ταραμπέλα. Δεν την ψηφίσαμε. Μπορούμε να την ψηφίσουμε ως προσθήκη. 171. Ως προσθήκη στη 41 υπέρ. Νομίζω χρειάζεται έλεγχο. 171. As Ως προσθήκη είπαμε. Πέρας ψηφοφορίας. Χάσατε. Απερίφημε μία ψήφο. Λοιπόν. Πού είμαστε τώρα. 177. Εψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν σας βλέπω τα χέρια. Είναι 42. Μα τι ψηφίσαμε, λέει ο κόσμος. Do not put to the vote, right. Amendment 43. Oh, no, they are adopted, yeah. Okay, fine. We vote 43. Right, we're just double checking all of this. 43. 43. Those in favor. Those against. Υπέρ κατά. Ε, εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επίσης. 45 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Υπέρ. Α, ας ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Έτσι. Την 180. Votes closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 147 λέει ο πρόεδρος. 47, όχι 100. Η 181 έχει αποσυρθεί. Ναι, αλλά είναι 47, όχι η 147 όπως λέει ο Πρόεδρος. So you have to vote on 47 now. Right. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 47. Παρακαλώ έτσι, να παρακολουθείτε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 182. με μια οριζόντια λέει τροπολογία που περιλαμβάνει είπε κατά ε, απορρίψετε η 48 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 50 είπε κατά και 49 Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί αυτές τις τρεις, 49, 50, 51. 49, 50 and 51. 49, 50, 51 είπε είπε... Εντάξει, εντάξει. Είναι πολύ περίπλοκο αυτό. Ψηφίζουμε τη 49, λοιπόν. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 50, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 51, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ωραία. Η συμβαστική 4, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τότε πάμε στην 53, την 188 και 89 μαζί. Υπέρ. Είναι προσθήκες. Κατά. Αποχές. 190 υπέρ. Υπέρ. Μάλλον χρειάζεται παλήθευση. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 190. On 90. The closed. Rejected. 50... Πέρας. Καταπίπτει. 54 ε, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 μέχρι και 58 μπορούμε μαζί. Οι δύο μεγάλες ομάδες είναι υπέρ. 55 μέχρι και 58 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική παριθμό 5 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά. Sorry. 61 in favor. Again. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 193, μάλλον κατά πίπτη, 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 δεν ψηφίζεται. 64 τα, τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 έχει αποσυρθεί 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπορούμε τις επόμενες μπλοκ, 67 μέχρι και 71 όλη τη σελίδα αν δεν διαφωνεί κανείς ωραία όλες μαζί τις ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται όλες. Η συμβαστική είναι 7 κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 και 74 ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 8 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.12 κατά πέφτει 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το παράρτημα τώρα το πρώτο καταπίπτει αν εγκριθεί η τροπολογία 1 2.15, 2.16 και 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 έχει αποσυρθεί, 221 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ, νομίζω αυτό χρειάζεται ηλεκτρονική απαλήθευση. 222 αρχίζει η ψηφοφορία. Votes Απερίφθη 15-19. 2-23 υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Abstentions, that's carried. Uh, 83 and 2... 83 και 24 υπέρ. Έλεγχος χρειάζεται και εδώ. Παρακαλώ 83 και 2-24 μαζί. vote is ah. Ah. Ah, Mr. is here. Έχει έρθει ο κύριος Κοφεράτη, όπως βλέπετε. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 15 κατά. 2,25 υπέρ. Κατά. Είπαμε ξανά. 2,25 υπέρ ψηφίζεται κατά. Οι φιλελεύθεροι ψηφίζουν. Αποχές εγκρίνεται. 2.26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 έχει ποσοστή 28-29. Α, όλη τη σελίδα μήπως μπορούμε να την ψηφίσουμε μαζί. Θα με υποχρεώσετε. μέχρι και τη συμβαστική 9, μέχρι την 90 στην άλλη σελίδα. Ε, υπέρ όλων αυτών είναι του εισηγητού οι Υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνονται όλες. Λοιπόν, και πάμε στη συμβαστική παρθμονενέα 9 με ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Απόχες εγκρίνεται. Ε, τώρα οι τελεγικές σκέψεις. Ε, η τροπολογία 92 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά. Απόχες απορρίπτεται. Η τροπολογία παρθούν 1 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 95 υπέρ. μάλλον θέλει έλεγχο αυτό. Για την 95 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρασα. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Και πάλι θέλει έλεγχο αυτό. Είναι μικρή διαφορά. Την 96 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μήπως άλλαξε κανείς γνώμη. Right. Well, their vote's closed. Πέρας. Απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά. Γι' αυτό το ελέγξαμε. 97. Υπέ Κατά. Α, και εδώ θέλει πολίτη. Παρακαλώ, 97 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. 97. No, 96 was rejected. Η 96 απερίφθη, οπότε ψηφίζουμε την 97. Πέρας. Απορρίπτεται. 97. Η τροπολογία 3 είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 6 έχει αποσυρθεί 103 υπέρ Α, θέλει έλεγχο 103 παρακαλώ ηλεκτρονικά That's closed. Εγκρίνεται. 18 υπέρ, 15 κατά. Η τροπολογία 7 και 104 μαζί ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 105 υπέρ. Υπέρ. Ξανά. Ας την εγκρίνουμε, ας την ελέγξουμε, συγγνώμη, την 105 ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι πέρασε. πέρασε. Ναι, εγκρίθηκε. Η 8 λοιπόν καταπίπτει. 106 είναι συμβατή με την 8 και με την 105. Ψηφίζουμε την 106 ηλεκτρονικά. Γιατί είναι τόσο μικρές διαφορές εδώ. Απερίφθη. Λοιπόν, η 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107 ως προσθήκη όμως, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 108 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται η 10 καταπίπτει 11 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται η 110 καταπίπτει 109 προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι 12 και 13 μπορούν να ψηφιστούν μαζί 12 και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 και 15 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 καταπίπτει 115 χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα το ζήτησε το ΕΛΚ αυτό τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ Α, εδώ θέλει επαλήθευση ηλεκτρονικά κατευθείαν για το δεύτερο τμήμα της 115. You Γιατί αλλάξατε γνώμη. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, το σύνολο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Το σύνολο, είπαμε όπως τροποποιήθηκε, πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα 35 υπέρ, κανείς κατά, μπράβο σας. Right. We're now going on to... Ωραία. Και τώρα, κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Έχουμε καθυστέρηση γρήγορα πρέπει να προχωρήσουμε. The draft opinion by Evelyn Gephardt. Σχέδιο γνωμοδότηση τη κυρία Gephardt ε, για τους λογαριασμούς πληρωμών. Πρέπει να ψηφίσουμε. Μήπως θέλετε κυρία Gephardt να πείτε τίποτε πριν αρχίσουμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα Βεβαίω να ευχαριστήσω θερμότατα τους και ηγητές μας. Το συζητήσαμε και χθες το βράδυ, είχαμε κρεμή ζητήματα και τα καταφέραμε όμως να τα διευκρινίσουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Υπήρξαν και κάποιες παρεξηγήσεις από ό,τι φαίνεται, τις οποίες καταφέραμε να ε, υπερβούμε και να ξεκαθαρίσουμε και μπορούμε να περάσουμε στην πληροφορία. Είναι πολύ σημαντικό ε, για τους καταναλωτές και την προστασία τους να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Good. All right. Right. Let's go then. Um, Μάλιστα, συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 82 πίπτη. Συμβιβαστική 15 κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Έναρξη ψηφοφορίας για το δεύτερο τμήμα. Uh, votes closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 17-16. 8 και 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την 85. Παρακαλώ ψηφίστε. Έχουμε αργήσει. Εγκρίνεται η 85. 86 υπέρ. Κατά. Έλεγχο, συγγνώμη, δεν είναι σαφές το πώς ψηφίζετε. Για την 86 μιλάω. Έναρξη 35 Τριάντα πέντε κάρτες. Ωραία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19-16. 9. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουν οι φιλελεύθεροι. Να το ελέγξουμε τότε. Γιατί είναι πολύ τσιμα τσιμα τώρα οι ψηφοφορίες. Λοιπόν. Πέρασε. Ε, έπρεπε, έπρεπε να, έρθει, να είχατε έρθει νωρίτερα αν θέλετε να μέτρηθεί η ψήφο σα. 87 κατά πίπτη, 88 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 13 τη εισηγήτριας υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 93 καταπίπτει. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. 98 υπέρ Καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Την 98. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας.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 Συγγνώμη, θέλετε έλεγχο τη 20? Ε, θέλετε να ελέγξουμε την 20. Ωραία. 20 λοιπόν. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σαφέστατα, όπως είχα πει. 107. Ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ έναρξη ψηφοφορίας για την 21 ηλεκτρονικός That's Εγκρίνεται. Μία ψήφος διαφορά. Ευτυχώς που το ελέγξαμε. 109. Συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Σηκώστε τα χεράκια. Καλά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικός. Την 110. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο ψήφοι διαφορά. 111. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Ψηφίζεται η φιλελεύθερη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παρακαλώ μου κάνετε ένα νόημα για τους, ε, από τους φιλελεύθερους να πάω πιο γρήγορα. Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 113. Υπέρ κατά τα αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 116 υπέρ κατά απορρίπτεται 117 υπέρ κατά Απορρίπτεται 118 υπέρ. Κατά. Α, απορρίπτεται 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 28 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 29 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 119 που είναι συμβατή με την 29, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 120 συμβατή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 121 υπέρ, Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 121 παρακαλώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. κατά. Υπέρ. να το ελέγξουμε καλύτερα. Την 126. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 18-18. Απορρίπτεται. 125. Υπέρ. Έναρξη ηλεκτρονικής πληροφορία για την 125. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κα... Υπέρ, υπέρ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 130 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος της 130 πέρας απορρίπτεται Συμβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 100, 38 συγγνώμη, υπέρ κατά εγκρίνεται 134 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 και 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά δύσκολο να πει κανεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα το 41 το ελέγχουμε ηλεκτρονικός. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά η 41. 42 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 του κύριου Ντεγιόγκ. Ένερξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. <coughs> Απορρίπτεται 18-18. 45 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικό 45. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 ψήφοι υπέρ. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 149 συμβατή υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Την 149. Πέρας. Απορρίπτεται 18-18. 150. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός, νομίζω ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έναρξη ψηφοφορίας στις 150 πέρας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτά λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη διορθώνει ο πρόεδρος. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε όλες αυτές να τις ψηφίσουμε μαζί αν μπλοκ. Διαφωνεί κανείς. 49, 50, 51, 52, 53, 54... Α, μέχρι την 53 λέτε. Καλά. Λοιπόν, 49 με 53. Τη κυρία Γέπχαρτ, υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνονται όλε 54. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Αυτή απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ Γιατί 57 μιλάω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 και 59 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 60 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ψηφίζουμε την την 61 ηλεκτρονικός. Τσίμα τσίμα θα είναι πάλι. Είναι. Απορρίπτεται μάλιστα. 18-18. 159. Υπέρ. Όχι, 161 διαμαρτυρίες ακούγονται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 καταπίπτει. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά Δεν είμαι σίγουρος. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς την 63. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά εγκρίνεται, σαφέστατα. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται επίσης. 67 ε, λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 68, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 69, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κα, υπέρ έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 3 Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 16 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και την τροπολογία 7 τελευταία υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης. Ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης Γκέπχαρτ. Πέρας. Εγκρίνεται. 33 ψήφοι υπέρ, 3 αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γκέπχαρτ. Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώνεται έτσι η ψηφοφορία μας για σήμερα. Κύριε Κοφεράτη, συγγνώμη. Γιατί θα σας τριμώξουμε λίγο χρονικά για τις δυο σας εκθέσεις. we ration some time on <laughs> So could I please ask you if you're not... Παρακαλώ πολύ, αν δεν ε, έχετε σκοπό να μείνετε, παρακαλώ όχι πολλές συζητήσει. I would like to, um, so... Λοιπόν, είμαστε λίγο στριμωγμένοι χρονικά. Είναι το επόμενο θέμα. Και θα ζητούσα από τους ε, σκιώδεις να είναι συνοπτικοί και λυτοί στις παρεμβάσεις τους. Την μεγάλη σημαντική έκθεση για τη διακυβέρνηση της ενής αγοράς σε σχέση με το εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο έχει το λόγο ο εισηγητής μας, ο κύριος Κοφεράτη, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς εδώ από την Επιτροπή πρώτα. Έχουμε. Θα μιλήσει για το θέμα αυτό. Καλώ ήρθατε κι εσεί που σα καθυστερήσαμε, συγγνώμη ζητώ. Η έκθεση για την διακυβέρνηση τη ενιαία αγορά κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξεταμίνου το 2014 το είχαμε συζητήσει για πολύ καιρό. Μα ενδιαφέρει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοφεράτη, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Η κυρία Γκάλπορτ είναι εδώ. Είναι εδώ. Ήταν εδώ. Ο κ. Μαρκάκης είναι εδώ. Κανείς από τους πράσινους. Εγώ είμαι εδώ για την ECR, ο κ. Διόγκ λείπει. Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος γιατί το θέμα το είχαμε συζητήσει και σε πρώτη συζήτηση. Χωρίς να επανέλθω στα ίδια θέματα, θέλω να κάνω κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις για το θέμα. Η σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι γνωστή σε όλους και το υπενθύμησε και ο Πρόεδρος νωρίτερα. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αυτός ο τρίτος πυλώνας που αφορά την ε, ενιαία αγορά διότι συμπληρώνει και τα οικονομικά θέματα και όσα είναι πιο στενά συνδεμένα με ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα ή απασχόλησης. Ο δεδηλωμένος στόχος, και επανέρχομαι στην πρώτε της μπροστά σας, ήταν να ορίσουμε το πλαίσιο και τα όρια του χαρακτήρα του τρίτου αυτού πυλώνα που συνδέει και αξιοποιεί και τους άλλους δύο επίσης. Εμείς πρέπει να στοχεύσουμε στο να ορίσουμε τις καθηγητήριες γραμμές αυτού που θα αποκαλούσαμε πραγματική οικονομία, ξεκινώντας από ορισμένου τομεί που είναι σημαντικοί για την ενιαία χώρα. Σημαντικοί για όλα, θεμελιώδους σημασίας θα έλεγα. Πρέπει να είναι υψηλή η συνοχή μεταξύ των διακεκριμένων σήμερα επιμέρους δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν κατόπιν σε μια σύνθεση όπως λέγαμε στο πλαίσιο του εξαμήνου. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε συνοχή από πλευρά ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να ζητήσουμε ωστόσο και το ίδιο να εφαρμόζεται και σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα πρέπει να έχει υπόψη της και να λαμβάνει υπόψη τον τρόπο προώθησης και την διαδικασία εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά δεν είναι μόνο κοινοτική πολιτική, είναι και πολιτική που εφαρμόζεται και από τα κράτη-μέλη ξέχωρα με σεβασμό της, νομισμό, της νομιμότητας και σύγκληση ως προς τους, τους στόχους. Στα μέσα Νοεμβρίου θα γίνει ετήσια ανάλυση για την ανάπτυξη, ιδίω δε θα εξεταστεί η έκθεση για το βαθμό υλοποίηση τη ενέας αγορά και άρα μια καλή ευκαιρία για έναν περαιτέρω έλεγχο της κατάσταση. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε από τη δημοσίευση αυτή θα μα είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Ο στόχος της δράσης, όπως έλεγα, έχει στόχο να εντοπίσουμε τα όρια του τρίτου πυλώνα και τον εντοπισμό βασικών τομέων. Γιατί ο τρίτος πυλώνας ορίζεται και στην έκθεση του κυρίου ΣΒΑΜ μεταξύ άλλων. Οι βασικοί κλάδοι πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια, η Επιτροπή δε να δώσει ενδείξεις που θεωρώ ότι παραμένουν σωστοί εμπολείς και να επιβεβαιωθούν. Είναι κλειδιά είναι οι υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η ψηφιακή αγορά. Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε και κάποια επιπλέον στοιχεία αξιολόγησης για την προστασία του καταναλωτή, των εργαζομένων και των πολιτών. Που ενδιαφέρονται από τις δραστηριότητε αυτών των κομβικών κλάδων. Γι' αυτό είναι σημαντικό θέμα η ανάδειξη και η επανακίνηση της βιομηχανικής πολιτικής. Δεν είναι αντικείμενο βέβαια της έκθεσης αυτής, αυτής αλλά ολόκληρης ενιαίας αγοράς. Το ίδιο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη τις δυνατότητες καινοτομίας και αύξησης γνώσης που προσφέρει. Κατόπιν, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ισχύ στο Single Market Act, όπου ήδη υπήρχαν θετικές απόψεις, ώστε ο κυκλικός, η κυκλικότητα και η μέθοδος που υιοθετούν να γίνουν κοινό τόπος κατά τη διάρκεια της περίοδου και να αφορά όλη την εσωτερική αγορά. Επίσης πρέπει να προβλέψουμε, να έχουμε στην εσωτερική αγορά καθορισμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών, δικαιωμάτων ιδιαίτερων, γιατί είναι ανάμεικτα με τα δικαιώματα ε, που σχετίζονται με την ε, οικονομική δραστηριότητα και την εργασία, ενώ αφετέρου με τα δικαιώματα του πολίτη. Κάτι τη διάρκεια της παρακολούθησης που θα κάνουμε στη διαδικασία αυτή και αυτό θα είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να δώσουμε νομοθετική περιγραφή στο θέμα αυτό σύντομα. Σε ό,τι αφορά το governance τώρα, πιστεύω ότι όταν καθορίζουμε τα όρια του governance πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση που, τις αναλύσεις που μας παρέχονται αλλά να μην περιοριζόμαστε όπως το έκανε η Επιτροπή σε πρώτη φάση, στην πρώτη προσέγγιση της ε, μιλώντας μόνο στην ποσοτική διάσταση. Είναι πολύ σημαντική η ποιοτική διάσταση ιδίως της υπηρεσίες αλλά και η αντίληψη της αποτελεσματικότητας που οι υπηρεσίες αυτές δημιουργούν στους πολίτες της Ένωσης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση σχέσεων μεταξύ πολιτών και υπό την, έννοια, υπό τη μορφή καταναλωτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε από αυτό το καθεστώς δυσαρέσκειας προσπαθώντας και από πλευράς μας εμείς να ενσωματώσουμε νομοθετικά τις απόψεις που στέλνουν οι πολίτες ως καταναλωτές αλλά και ως παραγωγή στους τομείς που μας ενδιαφέρει υπάρχει μια βελτίωση του ποσοστού ενσωμάτωσης των διατάξεων της εσωτερικής αγοράς από τα κράτη-μέλη. Θετικό, αλλά θα πρέπει να επιδιώκουμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Προφανώς. Αυτό είναι συνοπτικά οι συνοπτικέ θέσει μου. Ζητώ συγγνώμη γιατί μερικέ φορέ ήμουν πολύ απλουστευτικό, αλλά δεν υπάρχει χρόνο. Είμαι στη διάθεσή σα για τι περαιτέρω δραστηριότητε. Και εγώ μιλώ όχι μόνο για του σκιώδει ηγητέ, αλλά και για όποιον συνάδελφο θεωρεί ότι έχει παρατηρήσει που θα ήθελε να κάνει. Ευχαριστώ. Είμαι παραμένω στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ συνοπτική η έκθεση σωστά επιχειρήματα. Ο κύριο Σβάμπ νομίζω. Ο κύριο Σβάμπ. Μετά Χατζημαρκάκη, Ρούλε και βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να πω ειλικρινά ότι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη όχι μόνο για την περσινή ε, δουλειά που έτυχε να είμαι εγώ εισηγητή για αυτό το θέμα, αλλά γενικότερα για τη στόχευση, για την κατεύθυνση των επιχειρημάτων της προτάσεως που καταθέτει ο εισηγητής, είναι πάρα πολύ καλή. Όχι μόνο επειδή πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση με την περσινή πρόταση, αλλά και επί της ουσίας θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά τα όσα λέγει. Οπότε πιστεύω ότι φροντίζει και για τη συνέχεια των στόχων της έκθεσης και συνηγορεί προς την κατεύθυνση αυτή. Για την ε, έκθεση ε, για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να μας προβληματίσει αν η Ευρώπη χρειάζεται άραγε νέες αρμοδιότητες και εξουσίες ή μήπως αυτές που ήδη κατέχει να αξιοποιεί και εμείς να χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο τις εφιστάμενες δυνατότητες. Και σε αυτό καταλήγει και η έκθεση Κοφεράτη ότι δυστυχώς χωλένουν ακόμα κάποια πράγματα και υπολείπονται και αυτό θα πρέπει να γίνει απέτησή μας ευρύτατη πέρα από εθνικές αντιπροσωπίες και να την κάνει κτήμα της η Επιτροπή μας. Και είπα να είναι η σκιώδη μας η κυρία ε, γκάλ Πέλτς, όσο και αν μου στήχησε και είχα κάποια πικρία, ε, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντα οι ίδιοι που να ασχολούνται με ένα θέμα και ε, οριζόντια στο ευρωπαϊκό εξάμεινο να μπουν αυτές οι προτάσεις. Η πρόταση του κυρίου Κόφεράτη είναι πραγματικά απολύτως στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα βέβαια υπάρχουν μερικά σημεία που ήρθαν να προσθεθούν και έχουν να κάνουν και μέσα θέματα που βάζουν πάντα οι συνάδελφοι σοσιαλιστών και δημοκρατών δεν είναι κριτική προς την έκθεσή μα. Το βάζετε, το προτείνετε σε πολλέ εκθέσεις. Δεν αλλάζει τίποτα ε, στην ουσία και στην ποιότητα. Για τις συλλογικέ αγωγέ. ο, ο Επίτροπος Αλμούνια έκανε μια πρόταση, αλλά το ζητούμε σε τόσα χαρτιά μας. Δεν πειράζει να το ξαναφέρουμε και εδώ, δεν ε, χάλασε ο κόσμος. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια ενιαία και συνολική στρατηγική για την εξωτερική διάσταση πλέον της εσωτερικής αγοράς. Είτε αυτό θα γίνει με ελάχιστες προδιαγραφές, καλύτερα ή με το μέσο αμοιβαιότητας, θα το δούμε αυτό στην Ολομέλεια, στην ψηφοφορία. Αλλά από τη βασική κατεύθυνση είναι σωστό. Ε συμφωνώ. Κύριε Κοφεράτη, να πάρουμε επιτέλους τη μελέτη για το κόστος της μη Ευρώπης και να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα. Ζητώ και από τη Γραμματεία και από την Επιτροπή. Κανονικά ε, αναμενόταν η μελέτη να κατατεθεί στα τέλη της δικής μου εκθέσεως και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω τι απέγιναν αυτά τα σχέδια, αν εκδοκίμησαν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβαθύνουμε σε αυτή τη μελέτη, όπως λέγεται αυτό που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι πολύ τη μελετη οπως λεγεται αυτο που ανεθεσε η ευρωπαικη επιτροπη ειναι πολυ σημαντικο Χαίρομαι πάρα πολύ που η έκθεση αυτή, κύριε Κοφεράτη, διατρανώνει και πάλι ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν θα πρέπει να ε, προσανατολίζεται αμυγός σε μακροοικονομικούς παράγοντες που έχουν και αυτή τη σημασία τους, αλλά δεν μπορεί να είναι η αποκλειστική ε, για την αξιολόγηση μιας χώρας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε και επιγόντως ε, χώρες να μην πιέζονται ε, να κάνουν ε, διάφορες πολιτικές επιλογές λόγω οικονομικών δυσκολιών, αλλά να εφαρμόζουν παντού αποφάσεις που έχουν λάβει και εκείνα τα κράτη συμμετέχοντας στο Συμβούλιο, που έχουν συνδιαμορφώσει. Δηλαδή αυτό είναι στοιχειώδες στη δημοκρατία, να εφαρμόζονται οι λιμένες αποφάσεις χωρίς να επιβάλλεται τίποτα σε κανένα. Ε, χαίρομαι επίσης πάρα πολύ και θέλω να θυμίσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ε, τα όσα τους έχουν ε, ε, συστηθεί στα πλαίσια των συστάσεων χώρα, γιατί το έχουν συναποφασίσει και θα πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν τα έχει επιβάλει Τρόικα αυτά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν συναποφασιστεί, τα έχουν συνυπογράψει οι χώρες αυτά. Και πριν από λίγες εβδομάδες πάλι το ζήσαμε. Μας εκπλήσει αυτό. Οι χώρες δεν θέλουν να τους υπενθυμίζουμε πράγματα που έχουν υπογράψει. Μα δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι η Ευρώπη, ανεξαρτήτω ε, αρμοδιοτήτων εξουσιών περισσότερων ή όχι. Τα συμπεφωνημένα ισχύουν και εφαρμόζονται. γιατι οι συστάσει αναχώρα το είπα, να ενισχυθεί η αγορά και όχι μόνο τα μακροοικονομικά στοιχεία οπω είπαμε και τελο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, είναι καλή η έκθεσή του, θα γίνει καλή εν πάση περιπτώσει. Θέλω τη μελέτη αυτή που ζήτησε το Κοινοβούλιο σε βάθος για το κόστος της μη Ευρώπης, να το ξαναζητήσουμε για να έχουμε και καλύτερο και περισσότερο υλικό για τη συζήτηση και στις χώρες μας και που γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Χαντιμαρκάκης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφάρατη για την προεργασία του Πρέπει να πω ότι η έκθεση για μένα είναι υπερβολικά όριστη και γενική. Εντάξει, είναι γεγονός ότι επιτέλους χρειαζόμαστε ενιαία προσέγγιση, όπου η ενία αγορά να βλέπει και τις ε, ε, γενικότερες πολιτικές εξελίξεις της αγοράς και τις νομισματικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Καλό είναι αυτό, αλλά στα μέτρα που προτείνονται παραμένουμε υπερβολικά γενικόλογοι. Ε, δανείζομαι ένα μέτρο που προτείνει ο κύριος Κοφεράτη να έχουμε λιγότερες διαδικασίε προσφυγή επί παραλήψη και παραβίαση τη συνθήκη Το είπατε κι εσείς. Ναι, μπορώ να φανταστώ ότι αυτό έχει να κάνει ε, με τις προσφυγές που έχουν γίνει κατά της Ιταλίας. Εγώ ε, θέλω να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, και το είπε και ο κύριος Φαπ προηγουμένως. Αυτές οι διαδικασίες προσφυγής παραλήψης γίνονται για κάποιο λόγο. Διότι δεν επιτρέπεται να συμφωνούμε επί των αρχών, στην εκτέλεση να προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτές τις πολιτικές και να στρίβουμε δια του αραβόνος. Οι τρεις χώρες που είναι στην κορυφή της λίστας ε, αυτών των προσφυγών που είναι η Ισπανία, ε, Ιταλία πρώτη, Ισπανία και Ελλάδα αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι να αναφέρονται με το όνομά τους και να δημοσιεύονται κάποια στοιχεία, να προχωρήσει αυτό γιατί δεν μπορούμε εμείς να πάμε παρακάτω. Θέλω να το γυρίσω όμως, να μην αφήνουμε να μαστιγώνονται μόνο οι αμαρτωλές χώρες του Νότου. Να το γυρίσουμε ανάποδα. Είμαστε στο 20ο έτος της ενιαίας αγοράς και βλέπουμε την ψαλίδα να ανοίγει. Και αν δούμε το βαθμολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις επιδόσεις δηλαδή αναχώρα, κοιτάνε μόνο τι εφαρμόζεται. Δεν κοιτάνε όμως ε, τις σχέσεις που μπορεί να έχουν κάποια μέτρα με κάποια άλλα. Παράδειγμα, η Γερμανία στις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ε, ως κεντρικό μέρος της εσωτερικής αγοράς ε, είναι από τους πιο καλούς μαθητές αυτή τη στιγμή, αλλά απέχει πόρο από την υλοποίηση των στόχων στην έρευνα και την ανάπτυξη για να γίνει ένα άλμα ποιοτικό στην αλυσίδα παραγωγής. Γι' αυτό η Γερμανία μπλοκάρει τη θέση που θα μπορούσαν να πάρουν η Ισπανία, η Ιταλία ή η Ελλάδα. Μπλοκάρει λοιπόν την δυνατότητα ας πούμε, συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τον ανταγωνισμό για άλλες χώρες. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών του Νότου. Ισχύει αυτό. Γιατί το μπλοκάρει, λέει η κυρία ρούλε. Πώς δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ας πούμε, η Google, η Apple αυτού του κόσμου, οι μεγάλες εταιρείε <laughs> είναι στις Ηνωμένε Πολιτείε ή Samsung στην Κορέα. Αν δεν ε, επενδύεται ε, στην κορυφή, στην αιχμή του δόρατος, συνεχίζετε να είστε στην παραγωγή υποδέστερη. Ναι, αλλά πώς θα γίνει ότι αυτόματα θα μπουν οι άλλοι εκεί είναι ελπίδα, δεν συμβαίνει αυτόματα, αλλά ο συλλογισμό είναι αυτό. Ότι αν αυτοί που μπορούν δεν επενδύουν περισσότερο, πιέζουν και του άλλου προ τα κάτω. Τι εννοώ, θα πρέπει να έχουμε μια πανευρωπαϊκή αντίληψη. Η σημερινή σκέψη είναι βορρά-νότο. Δεν πάει έτσι όμω, θα πρέπει να δούμε και να μην λησμονούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ε, γιατί οι μεγάλες εταιρείες ε, λογισμικού που παραμένουν ακόμα στη Γερμανία όπως είναι η SAP σκέφτονται να σηκώθουν να φύγουν να πάνε στην Καλιφόρνια. Δηλαδή είναι και το εμπορικό ισοζύγιο των διαφόρων κρατών μεταξύ τους. Θα πρέπει να μπει στο σκόρμπορτο σε αυτό το βαθμολόγιο ή το, το πίνακα επιδόσεων. Δεν είναι καμιά τεράστια κατάκτηση επίτευγμα. Πρέπει να βελτιωθεί. Επόμενο θέμα που παραμένει γενικό λόγο ε, το θέμα της μετανάστευσης. Οικονομικά είναι σαφέστατο ότι τις χώρες που έχουν πλεόνασμα, που είναι οι χώρες του Βορρά αυτή τη στιγμή, αυτόματα προσελκύουν ένας μαγνήτης για ε, εργαζόμενους. Το ζούμε αυτό στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα. Νέοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ιταλοί και Έλληνες πηγαίνουν στην Αυστρία, Φιλανδία, Γερμανία. Εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί κανείς να το θεωρεί καλό, αλλά το συζητήσουμε ε, ανοιχτά και ειλικρινά. Αυτό που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη έλλειμμα είναι να υπάρχουν ε, μηχανισμοί ε, υποδοχής. Έρχονται οι νέοι που χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα στη Γερμανία και δεν βρίσκουν βοήθεια. Κάπου πρέπει να το δούμε και αυτό στην έκθεσή σας. Παραμένει και αυτό γενικόλογο. Θα κάνω και τροπολογίες αντίστοιχα προς τούτη την κατεύθυνση, έτσι ώστε το φαινόμενο αυτό να το αρπάξουμε από τα κέρατα ως άλλο τάβρο. Το ένα τελευταίο. Εδώ θα πρέπει να συζητούμε τέτοια θέματα, σε τούτη εδώ την Επιτροπή. Και όταν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτά για μένα είναι πολύ ε, περιορισμένα αυτά που προτείνετε Δημόσιες τράπεζες. Έχουμε αναπτυξιακές τράπεζες, όπως στη Γερμανία είναι η KFB, αλλά δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη τέτοιες. Ποιος θα μεταφέρει τα λεφτά στην πραγματική οικονομία, ποιος θα τα διαχειρίζεται. Χρειάζονται τράπεζες αναπτύξεως. Γι' αυτό εμείς φιλελεύθεροι θα κάνουμε ε, ειδική αναφορά σε τροπολογία. Τελευταίο, η ανεργία των νέων. Τι όφελος, ποιος ωφελείται από την ενιαία αγορά αν στην ε, Ισπανία είναι πάνω από 60% η ανεργία των νέων και στην Ελλάδα έχει φτάσει στο ρεκόρ του 70% και με μηνιαίους ε, ρυθμούς αυξάνεται. Εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε στην πολυθρόνα μας άνετα και βολικά. Πρέπει να βρούμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ένα σύμφωνο για την νεολαία, Youth Pact, θα μπορούσε να βοηθήσει αυτά τα στοιχεία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης να συμπεριλαμβάνονται και να βοηθούν για την αγορά εργασίας. Θα κάνουμε και εδώ τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Um, uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούλη. Θα είμαι σύντομη. Παρ' όλα αυτά όμως, ακριβώς λόγω του προλαλήσαντος θέλω να πω το εξής δεν είναι όλα τα θέματα δική μας αρμοδιότητα. Έχετε απολύτως δίκιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά αυτό λέγεται στην Επιτροπή Ήτρε. Και συζητείτε εκεί και στα άλλα έχετε δίκιο, αλλά στην ανεργία των νέων ε, ερχόμαστε στο παλιό θέμα. Είναι υποστήριξη των μικρομεσαίων. Και αυτό δεν με καλύπτει στην έκθεση. Ε, έβαλε τη βιομηχανία ο εισηγητή, ωραίο είναι αυτό και καλά, αλλά όταν αναφέρομαι στη βιομηχανία θα πρέπει τουλάχιστον να βάλω και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί βλέπω την ανάλυση σας και έχει μεγάλη σχέση με την ενέργεια των νέων. Αν υπάρχει εκπαίδευση, αυτή διτού τύπου με συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την κατάρτιση των νέων και θα παρακαλούσα τον εισηγητή να το γράψει και αυτό στην έκθεσή του. Γιατί έχω την αίσθηση ότι στην ευρωπαϊκή πολιτική και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι μικρομεσαίες ε, υμνούνται σε διάφορες ε, ε ομιλίες ε, και εξαγγελίες μεγαλόστομες, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, just... Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μερικά σχόλια, σχόλια ως σχέδιος εισηγητής. Καταρχάς θα συμφωνήσω με κάποια από τα σχόλια των συναδέλφων. Είναι μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σέργιο Κοφεράτη για αυτό αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα που έχουν να κάνουν ε, με την εσωτερική αγορά, κύριε Χατζημαρκάκη. Η διευκόλυνση για την ε, ε απασχόληση της ε, νεολαίας είναι, είναι αντικείμενο ξεχωριστής έκθεσης ε, που αφορά το εξάμεινο. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε παράλληλα με τα στοιχεία για την απασχόληση. Υπάρχουν τα στοιχεία της αγοράς. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε στα ζητήματα της ενιαίας αγοράς, να τα εμβαθύνουμε και να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Οπότε στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα απλώς να τονίσω σε σχέση με την κυκλική μέθοδο ε, υποβολής ε, πράξεων ε, για την ενιαία αγορά. Δύο φορές έγινε αυτό κύριε Κοφεράτη, ζητήσαμε και, και τρίτη αν θυμάστε, η οποία ε, δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ γιατί δεν τρελαίνεται για αυτή την ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο ελκυστική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρούμε ότι είναι ένας καλύτερος τρόπος ε, να πρωτοστατήσουμε ε, στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να δώσουμε πολιτική ε, έγκριση, να υπάρξει πολιτική έγκριση για κάτι τέτοιο. Αυτό που πρέπει όμως να σχολιάσουμε είναι συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένα στοιχεία. Στις οικονομικές εκθέσεις αναφέρονται συγκεκριμένα ε, στοιχεία βάσει συγκριτικής αξιολόγησης και ξέρω πολύ καλά ότι το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο ασχολείται και εκείνο με αυτό το θέμα, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση σε πληροφορίες ε, για το πώς θα πάνε οι αγορές στα διάφορα κράτη-μέλη και αν κάποια κράτη-μέλη δεν παίρνουν πολύ σοβαρά την ενιαία αγορά, αν έχουν καθυστερήσει στην εφαρμογή ε, της προστασίας των καταναλωτών, ε, την ενθάρρυνσή τους να είναι ενεργοί στην ε, ε, αγορά και τέτοιου είδους πράγματα. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν και να τα εξετάσουμε εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσουμε συγκεκριμένα και να ενισχύσουμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν ε, με την ψηφιακή ενία αγορά, γιατί αυτό έχει άμεση σχέση με την απασχόληση. Ένα πράγμα που θεωρώ ότι απουσιάζει και είναι σημαντική αυτή η απουσία από την έκθεσή σα και μου φαίνεται ότι είναι εξαιρετική σημασία. Είμαι σίγουρο ότι η κυρία Ρούλε θα συμφωνήσει. Οτιδήποτε για τι δημόσιε συμβάσει, οτιδήποτε έχουμε κάνει σε σχέση με τι μεταρρυθμίσει για το θέμα αυτό, για τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ύπαρξη ανταγωνιστικότερου περιβάλλοντο, τη καινοτομία. όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικοί δείκτες συγκριτική αξιολόγηση και απόδοση για την ενιαία αγορά και δεν τα βλέπω στην έκθεσή σα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε επικεντρωθούμε σε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε καλά και τα οποία κάνουμε καλά για να υπάρξει προστιθέμενη αξία στην έκθεση αυτή. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με το να συμπεριλάβουμε πολλά στοιχεία για τις οικονομικές υπηρεσίες που δεν αρμοδιότητά μας και αυτό το στοιχείο θα καλυφθεί από άλλες εκθέσεις. Ε, ίσως το καλό σας πλαίσιο να το χρησιμοποιήσουμε για την ενίσχυση πολλών άλλων πτυχών και να εξασφαλίσουμε βεβαίως ότι αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνουμε και αυτά ε, που συνεισφέρουμε στην ενιαία αγορά είναι σωστά. Για παράδειγμα, κινητικότητα, οικονομικές υπηρεσίες, ολοκλήρωση αυτών, ε, ε αξιολόγηση ομοτήμων, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να μην συνάδουν με τις διατάξεις ορισμένων τομέων της ενιαίας αγοράς. Εντάξει, αλλά πρέπει να ε, εστιαστούμε σε πράγματα τα οποία είναι αρμοδιότητά μας και τα οποία θέλουμε να βγουν ως αποτέλεσμα από αυτή την έκθεση. Μήπως μπορείτε να είστε λίγο ε, ε σύντομος κύριε Γκάλ ε, κυρία Γκάλ Πέτς για την τοποθέτησή σας γιατί έχουμε και άλλη μια έκθεση του κυρίου. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο να μιλήσω για το θέμα αυτό. Συμφωνώ με τις απόψεις του εισηγητή ότι ο συντονισμός ε, των πολιτικών απασχόλησης ε, και των οικονομικών πολιτικών θα πρέπει να συμπληρώνονται ε, και από άλλες παρεμβάσεις. Θα ήθελα καταρχά να πω ότι μπορώ να δεχθώ και να υποστηρίξω ως αφετηρία το πλαίσιο της έκθεσης αυτή. Είμαι πεπισμένη ότι αυτούς τους δύσκολους καιρούς μια σωστά λειτουργούσα εσωτερική αγορά είναι αναγκαία, καθότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς μπορεί να έχουν μόνο θετικές επιπτώσεις ε, στην ε, νομοθεσία εφόσον εφαρμόζονται σωστά και ενσωματώνονται σωστά από την εθνική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό δέχομαι ότι το έλλειμμα είναι σημαντικός παράγοντας, ωστόσο το αν είναι 0,6% όπως δείχνουν οι στατιστικές ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Ιδίω αν συμφωνούμε ότι αυτό ο τομέας είναι μέσο ουσιαστικό και σημαντικό για την πολιτική. Θέλω να τονίσω ωστόσο ότι δεν είναι σημαντικοί μόνο οι δείκτε, αλλά και η απευθείας ε, ποιοτικοί δείκτες σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση που είναι καλό, η έκθεση είναι ένα καλό πλαίσιο για να εξετάσουμε τους δείκτες αυτούς. Μπορώ να δεχθώ πλήρως την προσέγγιση του εισηγητή, να εξαρτάται η... να εμβαθυνθεί η δημοκρατική διαδικασία για τα εθνικά κοινοβούλια και να ενθαρρυνθεί ο ρόλος του ΕΚ. Είμαι βαθιά πεπισμένη ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε, ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια ε, προσέγγιση χωρίς διαφοροποίηση και συμφωνώ επίσης ε, με τον ε, ΣΥΓΙΤΗ, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η διαδικασία παραπομπής ε, είναι η μόνη λύση όταν καθυστερούν την ενσωμάτωση στα κρατημερικά. Την άποψή μου πρέπει να προχωρήσουμε με τις ενημερώσεις, τακτικές ενημερώσεις επιτροπής για το περιεχόμενο των, της νομοθεσίας. Κάτι άλλο που θεωρώ είναι ότι για να προωθηθεί ο διάλογος και να μάθουμε από την εμπειρία επιτόπου θα πρέπει να ενισχύσουμε στο φόρουμ, το φόρουμ αυτό τώρα. Τελει σημαντική, βασική παράγοντες. Συμφωνώ με τις απόψεις του κ. Κοφεράτη ότι είναι αναγκαίο να έχουμε μια ενοποιημένη βιομηχανική πολιτική για την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών και για να οικοδομήσουμε, να βγούμε με σταθερό τρόπο από την κρίση. Πιστεύω ότι είπα τα πάντα Ήμουνα σύντομη, προσπάθησα να καλύψω πολλά σημαντικά θέματα, περιμένω σε μια συνεργασία με τους ε, συναδέλφους και ευχαριστώ τον πρόεδρο που μου έδωσε το λόγο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχει το λόγο όμως η εκπρόσωπος της για να πει δύο πράγματα. Και μετά ο κ. Σκοφεράτη να συνοψίσει. Σας ε, Πι, πιέσαμε πολύ κύριε Κοφεράτη, συγγνώμη γι' αυτό. Κύριε Βεχόβεν, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτον, και εγώ θα είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που δώσατε στο να μετατρέψουμε την ενιαία αγορά σε ένα βασικό, μια βασική παράμετρο του, εξαμή, του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Εμείς εξετάσαμε με την έκθεση που εκδώσαμε πέρυσι την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε βασικούς παράγοντες και σε βασικά σημεία της, των κρατών μελών. Φέτος θα ετοιμάσουμε ο Σονούπο στις 30 Νοεμβρίου μια δεύτερη έκθεση ενσωμάτωσης μπαίνοντας σε περισσότερες λεπτομέρειες βλέποντας πού είναι τα κενά, ποια προβλήματα υπάρχουν και πού έχει επιτευχθεί πρόοδος για να μπορέσει η ενιαία αγορά να δουλέψει καλύτερα, να παράσχει περισσότερα. Ευχαριστούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο για τη βοήθειά σας να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, φέτος για πρώτη φορά ετοιμάσαμε το δικό μας scoreboard βαθμολόγιο των κυβερνήσεων που περιέχει ωστόσο και προσπάθειές μας να ε, χρησιμοποιήσουμε την, τα αριθμητικά στοιχεία όταν κάνουμε μια πιο ποιοτική ανάλυση της πορείας προς την ενιαία αγορά, ούτως ώστε να έχουμε πιο τεκμηριωμένα ε, δεδομένα αργότερα. Για τους βασικούς τομείς χαίρο που βλέπω ότι όλοι υποστηρίζετε τις θέσεις μας εκεί. Οι βασικοί τομείς είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να εξετάζουμε και συμφωνούμε με τους τομείς που ανέφερε ο εισηγητής. Και δύο λόγια ακόμα για να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας συνολικά σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι συμφωνούμε πως αν θέλουμε να βελτιωθεί η ενιαία αγορά θα πρέπει να δουλέψουμε σε, σε μια σειρά τομέων για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή ενσωμάτωση. Μας, ικανοποιεί, οι, μας ικανοποιούν οι βελτιώσεις που βλέπουμε εδώ, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ λοιπόν για την έμφαση που δίνεται στις δικέ μα προτεραιότητε και γιατί συνεχίζει να ασχολείστε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί με πολύ χαρά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σα σε σχέση με όλα αυτά που αναφέρατε. Κύριε Κοφεράτη, μπορείτε να συνοψίσετε και να μα πείτε για το χρονοδιάγραμμα. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ καλή θα τα πω γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Πρώτον, ευχαριστώ για τι παρατηρήσει. Κάποιες από αυτές είναι πολύ σημαντικές, αλλά αποτελούν τμήμα της κατάστασης των συζητήσεων. Είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε γενικά θέματα τώρα. Προφανώς θα αρχίσουμε να χτενίζουμε τα κείμενα αργότερα, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από γενικές συνολικές παρατηρήσεις για να φτάσουμε σε λεπτομέρειες κατόπιν. Κάποιες από τις παρατηρήσεις είναι πολύ χρήσιμες. Θύμισε ο πρόεδρος και τον ευχαριστώ γι' αυτό για τις δημόσιες προμήθειες και αυτό πρέπει να ενταχθεί στην έκθεση γιατί είναι και μια δουλειά που μαζί κάναμε και που είχε μια πολύ θετική έκβαση. Πού θα, πότε θα τελειώσει είναι άλλο θέμα. Να πω στον κύριο Χατζημαρκάκη να μην ανησυχεί σε ό,τι αφορά τις γενικές αναφορές. Εμείς στις λεπτομερίες θα μπούμε στο κείμενο θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά σε κάποια σημεία πρέπει να παραμείνουμε γενικοί, γιατί μιλάμε για την ενιαία αγορά. Υπάρχουν τομείς που ανήκουν σε άλλες οδηγίες και άρα σε άλλες επιτροπές, που κάνουμε παραπομπές γενικού χαρακτήρα μόνο. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε υφαρπάζοντα τη δουλειά που κάνουν άλλες ή που πρέπει να κάνουν άλλες επιτροπέ. Ό,τι αφορά την αναφορά στι διαδικασίε παραπομπή, μην υπάρχει παρανόηση. Εγώ δεν το έγραψα διότι θέλω να δοθεί α πούμε άφησε μαρτιών στη χώρα μου. Έχει σοβαρέ ευθύνες η Ιταλία διότι ένας κανόνας που, που υιοθετείται εδώ πρέπει να ενσωματώνεται. Αν δεν ενσωματώνεται υπάρχουν τιμωρίες. Αυτό που είπα είναι να γίνονται συζητήσεις περισσότερες εδώ. Όχι να αλλάζουμε αφού εγκριθεί ένας νόμος. Εγώ έκανα μία, ένα σχόλιο και μην νομίζετε ότι κρύβεται πίσω από αυτό ότι είμαι, θέλω να είμαι επίοικης κατά των κακών μαθητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. για το χρονοδιάγραμμα Τροπολογίε μέχρι τι 25 Νοεμβρίου 12 η ώρα το μεσημέρι. 16 και 17 θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. συμβαστικέ 9, συμβαστικές 9 Ιανουαρίου και θα εγκρίνουμε στις 23 Ιανουαρίου για να πάμε ε, στην Ολομέλεια μαζί με την Επιτροπή Οικονομικών και Ασχόλησης ε, το Φεβρουάριο του 2014. Αυτό είναι το χρονοδιαγραμμά μα. Θα είναι ένα σημαντικό τμήμα το να ε, τεθεί και πάλι η προώθηση της ενιαίας αγοράς ε, στο επίκεντρο. Συγγνώμη, κύριε Κοφεράτη, που ε, σας τριμώχνουμε λιγάκι. Μήπως μπορείτε να είστε λίγο σύντομο σε σχέση με τις τροπολογίες. Από ό,τι βλέπω γύρω στις 60 ήταν. Ας ακούσουμε τώρα την άποψή σας και μετά μπορούμε να κάνουμε τη συνάντηση με τους κύριους συζητητές Κρόιτσμαν και Σφάμπ, ο οποίος κύριος Σφάμπ αντικαθιστά και την κυρία Πιετικάινεν, η κυρία Ρούλε δεν είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Δεν είναι πολύ λοιπόν από τους κοιόδους συζητητές σας εδώ. Παρ' όλα αυτά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η απόψή σας για τις τροπολογίες. Μπορείτε να μας κάνετε ένα σύντομο σχόλιο. Ποια είναι η αντίδρασή σας σε σχέση με τις τροπολογίες. Ναι, είναι χρήσιμη η ένδειξη αυτή γιατί μπορεί να υπάρξουν δυσκολίε ό,τι αφορά την συζήτηση που θα κάνουμε σε πολύ περιορισμένο χρόνο. Μπορεί να παρακάμψουμε πολλά πράγματα με μια συνάντηση σκιωδών που μπορεί να αντιμετωπίσει το ό,τι θέμα δεν θα μπορέσει να συζητηθεί εδώ. Την άλλη εβδομάδα θα σας στείλω, προτίθεμαι να σας στείλω, συνθετικές προτάσεις. Άρα θα έχετε σύντομα τα συμβιβαστικά κείμενα στη διάθεσή σα. Και αυτό θα είναι και μια περαιτέρω ευκαιρία να τα δούμε πιο λεπτομεριακά μαζί με αυτά τη ε, γενικότερης συζήτησης. Τα θέματα που συζητήθηκαν στην έκθεση και ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που κάνετε και τις ε, προτάσεις ε, ενίσχυσης. Ένα από τα κύρια θέματα πάντως και η σύνθεση εδώ θα είναι εύκολη, διότι δεν είναι εύκολο να τα αναφέρουμε όλα, αφορά τις καθηγητές γραμμές για τις επιχειρήσεις. Όλοι συμφωνούμε ότι οι γραμμές αυτές πρέπει να θεσπιστούν, η μη ή το έργο που θα κληθούν ε, να κάνουν επιχειρήσεις, δεν θα έχει αποτελεσματικότητα. Πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας την πρόταση που θα σας κάνω Ελπίζω να είναι αποτελεσματικά και αυτό που ζητώ από σας είναι να μου δώσετε ιδέες που δεν θα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις γιατί δεν πρόκειται να το εφαρμόσουν αλλά που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους και θα έχουν εγκάρσια επίδραση στην έκθεση. Πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε η διαφάνεια, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει μεγαλύτερη ορατότητα των επιχειρήσεων να είναι να αναδεικνύεται και όχι το ανάποδο, δηλαδή να μην δημιουργείται δημιουργούνται δυσκολίες σε κάθε επιχείρηση που θα υπάγονται στη διαδικασία αυτή. Είναι σημαντικό να έχουμε μία θετική θέση στην ενσωμάτωση από χώρα σε χώρα. Εκτίμησε επίσης και τις τροπολογίες για την εμπλοκή ορκωτών λογιστών που γνωρίζουν καλά την ρητή ανάλυση των θεμάτων που ρυθμίζονται από την οδηγία. Θα πρέπει, όπως το ζητούν και κάποιες τροπολογίες, να προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους και το χρόνο εμπλοκής των ενώσεων εργαζομένων. Το θέμα των stakeholders είναι σημαντικό. Και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις διαφορές που υπάρχουν. Κάποιες τροπολογίες του συναδέλφου Κρόιτσμαν, ε, δεν με πείθουν, το λέω με ειλικρίνεια. Διότι μπορεί και αν κατάλαβα λάθος. Και αν κατάλαβα λάθος, να αλλάξω την άποψή μου ενδέχεται να καταστήσουν στην ουσία προαιρετικό το θέμα επιλογής επιχειρήσεων ή να μειώσουν σημαντικά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εισαγωγή του νομοθετικού αυτού κειμένου. Το είπα και νωρίτερα ότι η ιδέα του να δουλέψουμε για κάτι που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να υποστούν μεγαλύτερο κόστος δεν πρέπει να είναι ο στόχος μας. Από την άλλη δεν πρέπει να μπούμε στην περιπέτεια της περιγραφής κανόνων που κατόπιν θα αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί και θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να απομακρυνθούν από τις επιταγές που θέλουμε να τους επιβάλλουμε. Αυτά είπα ότι είμαι διατεθειμένος όχι μόνο να σας ακούσω αλλά και να κάνω αν χρειαστεί και μια άλλη συνάντηση για να μπορέσουν οι σκιώδεις να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Όταν την άλλη εβδομάδα σας στείλω τα κείμενα, τα συμβιβαστικά. Um, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο για σύντομα σχόλια. Από τους κύριους συζητητές. Κύριε Σφαπ, θέλετε? Όχι. Κύριε Κρόετσμαν τότε. Αναφέρθηκαν ήδη οι τροπολογίες σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ Μάλκομ. Εγώ ε, μένω όμως. Στην πρώτη συζήτηση με... Ε, ε, αντικατέστησε ε, και αντιπροσώπησε ο κύριος Χατζημαρκάκης. Εγώ έχω επί της αρχής προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βγαίνουν και βγάζουν ωραίους λόγους τις Κυριακές στα μπαλκόνια να μειωθεί η γραφειοκρατία για το ένα και το άλλο. Και έρχεται η Δευτέρα και κάνουμε μια πρόταση που σημαίνει 42.000 επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη ενέχονται, δηλαδή τις αφορά. Το είπα και παρουσία του Επιτρόπου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο ε, χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, στο DAX και τα λοιπά, το έχουν ως προπαγάνδα χρησιμοποίηση αυτό. Και γιατί να μην το κάνουν και μικρές επιχειρήσεις. Ε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Το πολύ πολύ εθελούσια ε, ρύθμιση. Ε, και ε, κοιτώντας τις τροπολογίες φοβούμε ότι ε, επιφορτίζουμε τις επιχειρήσεις με πλέον γραφειοκρατία και είναι και επικίνδυνο να πάμε στους 250 εργαζομένους σε αντίθεση με τις 500. Το αντίθετο συμβαίνει. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε και να σώσουμε τις ε, μικρομεσαίες, τελικά να διπλασιάσουμε, όχι να μειώσουμε στο μισό είναι υπερβολική αυτή η επιβάρηση. Δεν έχουν μεγάλα τμήματα και υπηρεσίες να ασχολούνται με αυτά. Το έχω πει και την περασμένη φορά. Πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα αυτά, να ενοποιούνται, να ελέγχονται και πάει λέγοντας. Και το κόστος δεν είναι μόνο για την ίδια την εταιρεία, έχει και παρεπόμενο κόστος. Έχει μεγαλύτερο νόημα αυτό που πρότεινε ο κύριος ε, Χάρπορ να περιοριστούμε στις εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείες. Γιατί γι' αυτό ενδιαφέρονται κυρίως οι επενδυτέ και η κοινή γνώμη. Τώρα για τις μικρομεσαίες όχι. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για κάθε επιχείρηση να αποφασίζει ε, που θα συμμετέχουν. Υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις ε, και ε, μέτρα που προσφέρονται περισσότερο για κάποιες εταιρείες ή για κάποιες χώρες. Εντάξει, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά όχι δεσμευτικές, να μπορούν να επιλέγουν οι επιχειρήσεις και να τους βοηθούμε. Αυτό που προτείνεται δεν είναι αυτό. Δημιουργούμε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη, ένα επιπλέον. Αφήστε δε πω αυτό, το CSA αφορά εταιρείε που δραστηριοποιούνται διεθνώς και θα πρέπει να λογοδοτούν. Γενικά είμαι αντίθετος και η ανάλυση του κινδύνου ε, ουσιαστικά τιμωρείται. Τι είναι αυτό. Υπάρχουν τομείς όπου αυτό το CSR έχει νόημα. Το πώς θα αποφασιστεί δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση για το πώς θα λειτουργούν οι εταιρείε στο εσωτερικό του. Και η πρόταση ένα χώρα country by country, είναι κάτι ε, που θεωρώ ότι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της προτάσης. Και τέλος, ε, θα ήθελα να πω κάτι για αυτό που προτείνουν ορισμένοι συνάδελφοι. Υποχρέωση δημοσίευσης σε όλη την αλυσίδα των προμηθευτών. Μα ήδη από τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν τελείως αναδαφικά αυτά που ζητούσανε. Και τώρα και τους προμηθευτές να βάλουμε μέσα, ωραία. Εκεί να δείτε επιπλέον κόστος. Και δεν είναι μόνο για τις ε, ε, επιχειρήσεις και για ε, εκείνους που τους προμηθεύουν. Δεν ξέρω αυτό, όπως θέλετε να το φανταστείτε, να το υλοποιείτε στην πράξη. Να αφήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις να λειτουργούν με την ησυχία τους και χωρίς υπερβολική επιβάρυνση και υπερβολικό κόστος. Αλλιώς λέμε για την ανταγωνιστικότητα, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και φέρνουμε τη μία πρόταση μετά την άλλη που έχει επιπλέον κόστος, χωρίς να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα. Και το λέω πολύ συνειδητά αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κρόιτσμαν. Αναφερθήκατε και στι δικέ μου τροπολογίε Προσπάθησα να ευθυγραμμιστώ κάπως με την κατεύθυνση που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το πεδίο εφαρμογής αυτού του πράγματος να ε, αναφέρεται κυρίως, στην ε, ε, υποβολή εκθέσεων στους μετόχους. Πρέπει να πάμε προς κάποια κοινά, προς κάποιες κοινέ προδιαγραφές που πρέπει ακόμη να αναπτυχθούν βεβαίως. Είναι μια πρόταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για την αναθεώρηση των οδηγιών περί ε, λογιστικών της τέταρτης και της έβδομης οδηγίας. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αρκετά επίπονη και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην περιορίσουμε υπερβολικά τα πράγματα, να είναι και σαφές το νομικό πλαίσιο των επιχειρήσεων Υπάρχουν κάποια στοιχεία τέλο πάντων για τα οποία πρέπει κάπως ε, να δουλέψουμε. Θα ήταν χρήσιμο να συνεργαστούμε με τον κύριο Κοφεράτη. Θα μας στείλετε ούτω ή άλλω συμβιβαστικέ τροπολογίες, οπότε θα μας δώσετε ένα πλαίσιο συζήτησης. Είναι εδώ κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσατε βέβαια πολύ προσεκτικά. Θέλετε να μας ενημερώσετε σχετικά ή όχι για το θέμα του κυρίου Μπαλτασάρη, μήπως μπορεί κανείς να μας ε, ενημερώσει. Ένας θόρυβος ακούγεται. Α, σταμάτησε. Okay, all right. Μάλιστα. Τότε κάποια άλλη στιγμή θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή θέλετε τελικά να πάρετε το λόγο πριν ε, ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα σχόλια. Εξετάσαμε τις τροπολογίες αυτές. Περιμένουμε τώρα την οριστική έκθεση της Επιτροπής ΥΜΚΟ. Μάλιστα. Κάποιο έχει κάπου ένα ανοιχτό μικρόφωνο και δημιουργείται ένα πρόβλημα με τα μικρόφωνα γενικώ. Α, όχι, ξανάρχισα. Α, είναι απ' έξω θόρυβο. Καλώ. Κύριε Κοφεράτη, θέλετε τότε να συνοψίσετε ή να μας πείτε για το χρονοδιάγραμμα. Προτείνουμε 28 Νοεμβρίου να ψηφίσουμε. Ε, θέλετε να συμφωνήσετε με αυτό, να διαφωνήσετε, υπάρχουν ε, άλλα σχόλια. Μια γενική παρατήρηση. Καταλαβαίνω mm. τις αμφιβολίες ε, και τις επιφυλάξεις που εξέφαζε ο κ. Κρόιτσμαν και εσείς πρόεδρε. Πρόκειται για αντιρρήσεις που προέρχονται από μια καθόλου σεβαστή φιλελεύθερη προέλευση. Πρέπει να βρούμε ένα σημείο σύγκλησης. Θα ήθελα να είχαμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε τι είναι πιο αποτελεσματικό σήμερα για μια επιχείρηση. Η απελευθέρωση από τους δεσμούς και η υποταγή σε μια αγορά που την ε, συνθλίβει ή να είναι στα πλαίσια μιας ελεγχόμενη αγορά που κατόπιν τη επιτρέπει ωστόσο να απελευθερωθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τη συζήτηση, σε άλλο πλαίσιο θα γίνει και θα μιλήσουμε μετά την υποβολή των συμβαστικών τροπολογιών συζητώντα την δυνατότητα να τα βρούμε. Αυτά. Και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πολύ γρήγορα μας παρουσιάσετε δύο ε, εκθέσεις. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς που έμειναν λίγο παραπάνω. 3.30 θα αρχίσουμε σήμερα το απόγευμα γιατί υπάρχει μια ε, ειδική διάσκεψη των ε, προέδρων και θα έχουμε μια ακρόαση για τα οργανωμένα ταξίδια μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα μετά ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο e-call. Οπότε με χαρά θα, τα, θα σας ξανασυναντήσω το απόγευμα στις 3.30. Ευχαριστώ.